Good morning, colleagues. Mrs. Hennis, I love your backpack. <laughs> Good morning. <laughs> Um, I apologize for the... Ζητώ συγγνώμη γιατί καθυστερήσαμε λιγάκι. Σήμερα θα συζητήσουμε τις ε, επιπτώσεις της συνθήκης της ε, Λισαβόνας ως προς την ε, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη μετά από τη θέση σε ισχύ της ε, νέας συνθήκης και μετά θα γίνει μια συζήτηση για το SWIFT και PNR ε, υπό την παρουσία του κυρίου Τζόναθαν Φόλ, ο οποίος θα ε, φτάσει στις 10 από ό,τι μου είπαν. Προτείνω λοιπόν να αρχίσουμε άμεσα. Όπως γνωρίζετε, εργαζόμαστε από χτες υπό νέο καθεστώς και σήμερα θα δούμε τι επιπτώσεις θα υπάρχουν ιδιαίτερα ως προς τον νέο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διεθνείς συμφωνίες, δύο εκ των οποίων ήδη ανέφερα, καθώς ε, και τις επιπτώσεις ε, της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η οποία είναι ε, δεσμευτική, νομικά αν δεν ξέρω πώς και πώς θα έχουν τα opt-outs, οι αυτό Θα δώσω όμως το λόγο στον κύριο Πάσος της νομικής υπηρεσίας ο οποίος ε, μας έστειλε ένα υπόμνημα με ορισμένα σημεία. Κύριε Πάσος, θα ήθελα να μας κάνετε μία σύντομη εισήγηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, όπως είπατε. Σας ε, έχω δώσει μία σκιαγράφηση που ίσως θα διευκολύνει τις σημερινές συζητήσεις. Ήλπιζα να κάνω την παρουσίαση σε τρία μέρη. Καταρχήν που προερχόμαστε, από πού προερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Δηλαδή ε, σε σχέση με τη συνθήκη της Νίκαιας και τη συνθήκη της Λισαβόνας. Το δεύτερο τμήμα αφορά την τρέχουσα κατάσταση ως προς συμφωνίες που υπεγράφησαν από το Συμβούλιο. Um, Και εάν νομίζετε ότι έχουμε χρόνο, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την δράση της Επιτροπής στο μέλλον σε σχέση με τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών γενικότερα. Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν ε, είναι ανάγκη να μπω σε λεπτομέρειες για, τις, ε, για τη διάταξη του άρθρου 24, τη συνθήκη της νίκης και το τι έχετε στα χέρια σας τώρα. Είχατε μία διακυβερνητική διάρθρωση για τον τομέα των ελευθεριών, ασφάλειας και δικαιοσύνης με μία διάταξη η οποία συνδεόταν με το CFSP, με την ΚΕΠΑ. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κοινοτική μέθοδο ως προς την, ε, το ρόλο του Συμβουλίου καθώς και της ε, Επιτροπής που μπορεί να υποβοηθήσει τη δάση του Συμβουλίου. Άρα δεν υπάρχει δικαιοδοτικός έλεγχος από το Κοινοβούλιο. Το τελευταίο στοιχείο είναι η δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να εκφράσουν εθνική επιφύλαξη η οποία έχει εκφραστεί πολλές φορές ιδιαίτερα σε σχέση με το PNR όπου 11 κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν την δυνατότητα του άρθρου 24 παραγράφου 5 το οποίο σημαίνει ότι η προσωρινή εφαρμογή μπορεί να ισχύσει, δηλαδή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν τη συμφωνία, η οποία βεβαίως είναι κάπως ε, προβληματική. Τώρα έχουμε νομική προσωπικότητα, νομικό πρόσωπο, άρθρο 47, ειδική πλειοψηφία επίσης στο Συμβούλιο ως γενικό κανόνα θα δρούμε με βάση τη συναπόφαση. Το ενδιαφέρον με τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι ότι έχουμε μία και μοναδική ε, διάταξη για τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών και την ε, συμφωνία, τη σχετική συμφωνία και σύναψή του σε σχέση με τις συμφωνίες ΚΕΠΑ άρθρο 218 το οποίο φέρει λεπτομέρειες για το τι κάνει το Συμβούλιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων, υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή, ποιος είναι ο βασικός διαπραγματευτής, ποια είναι η ομάδα διαπραγματευτών και βεβαίως ο, ο βασικός διαπραγματευτής είναι η Κομισιόν εκτός και εάν έχουμε την ύπατο εκπρόσωπο και αυτό που έχει, σημαντικό, που έχει σημασία για την Επιτροπή σα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία κάθε φορά που υπογράφεται μια διεθνή συμφωνία από το Συμβούλιο, διότι υπάρχει η συναπόφαση και ε, το άρθρο 218.6BA λέει ότι χρησιμοποιούμε την κανονική ε, νομοθετική διαδικασία ως προς ελευθερίες, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Ως προς το θέμα που σας ενδιαφέρει πιο άμεσα, α, είναι η, τι γίνεται με τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, μάλλον που έχουν τύχει διαπραγμάτευση αλλά δεν έχουν συναυθεί. Αν ε, δεν είχε κάτι τέτοιο δεν θα το συζητούσαμε καν. Αλλά τη στιγμή που έχουν καταρχήν υπογραφεί θα πρέπει να τα εντάξουμε όλα στη συνθήκη της Λισαβόνας, δηλαδή τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτή τη διάταξη, δηλαδή το 2018 θα ισχύσει. Επίσης θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ υπογραφής και θέσης σε ισχύ, διότι η υπογραφή δεν δεσμεύει νομικά. Ακολουθούμε τη σύμβαση της Βιέννης Πρόκειται για μια συμφωνία επί ενός κειμένου από τα συμβολόμενα μέρη και τα συμβαλόμενα ε, μέρη δεν θα πρέπει να παραβούν τη συνθήκη, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι η υπογραφή δεν σημαίνει ότι δεσμεύονται τα συμβαλόμενα μέρη. Χρειάζεται κύρωση ή σύναψη που είναι η λέξη που, χρησιμοποιούμε, που χρησιμοποιούν συνθήκες. Όλες αυτές οι συμφωνίες λοιπόν που έχουν υπογραφεί και είναι επτά αυτές Άρα τώρα το Συμβούλιο θα πρέπει να ζητήσει τη συνένεση του Κοινοβουλίου. Η συνένεση είναι η σωστή διαδικασία, άρα τώρα θα πρέπει να ζητήσουμε μία επιστολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντας τη συνένεση. Αυτό αυτό δεν αφορά διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου, είναι ε, νομική υποχρέωση και το Συμβούλιο δεν πρέπει να ε, μακροχρονίσει, διότι θα πρέπει να ζητήσει την ε, συνεργασία του Κοινοβουλίου και το Κοινοβούλιο αναμένει κάτι τέτοιο από το Συμβούλιο. Και τώρα έχετε δύο δυνατότητες. Τη στιγμή που έχετε την επιστολή από το Συμβούλιο ζητώντας τη συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. είτε συνενεί το Συμβούλιο με τη συμφωνία που έχει υπογραφεί, άρα θα τεθεί σε ισχύ, θα κυρωθεί και θα τεθεί σε ισχύ και θα δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε το Κοινοβούλιο δεν συνενεί με τη συμφωνία όπως έχει υπογραφεί. Και τώρα το ζήτημα είναι, σε αυτή την περίπτωση μπορεί η Επιτροπή αυτή ή το Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Επιτροπή να επαναδιαπραγματευτεί. απάντηση είναι αρνητική, διότι η συμφωνία έχει υπογραφεί, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες να ξανανοίξουν δηλαδή οι διαπραγματεύσεις. Δηλαδή είτε συνενούμε είτε όχι. Εάν όχι, τότε δεν μπορεί να συναυθεί η συμφωνία και δεν θα έχει νομικές, νομικό αποτέλεσμα. Άρα η Επιτροπή θα πρέπει να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση εδώ. Δεν υπάρχει πια η Προεδρία του Συμβουλίου, έχουμε την Κομισιόν πλέον και η Κομισιόν θα προτείνει στο Συμβούλιο την ε, ε, πρόταση συμφωνίας ή την πρόταση απόφασης. Ως προς, την, ε, όπως προς συμφωνίες που έχουν την που ε, υπάγονται σε αυτή την υποχρέωση, εάν δεν συνενέσει η Επιτροπή, τότε δεν λήγουν οι προσωρινές υποχρεώσεις. Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 25 της Σύμβασης της Βιέννης, εάν ένα συμβαλόμενο μέρος δεν θέλει να συνάψει συμφωνία, τότε δεν ισχύει η προσωρινή εφαρμογή. Επίσης, όλες αυτές οι διαδικασίες που ίσχυαν δυνάμει του 24-5 για τις εκκρεμείς συμφωνίες δεν ισχύουν, εκπίπτουν διότι η νομική βάση έχει καταργηθεί. Και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για την ειδική κατάσταση ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Δανία, αλλά θα πρέπει να ισχύσουν τα πρωτόκολλα 21 και 22. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα για 2-3 λεπτά να σας πω πώς διαβλέπουμε το μέλλον και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τώρα που έχουμε την ε, μεγάλη αυτή συνένεση που σημαίνει δραστική αλλαγή για την ε, δική σας Επιτροπή και ως προς την Επιτροπή Αλληλείας που είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα τώρα χρειάζεται συνένεση και ίσως θα πρέπει να δούμε, να ζητήσουμε δηλαδή ε, τη συνένεση κάτω από όλες τις συνθήκες. Στο άρθρο 2.18, παράγραφος 2, που είναι η βασική διάταξη για τη διαπραγμάτευση σύναψη συμφωνιών, το Συμβούλιο ορίζει την εντολή των διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν έχει αλλάξει και με βάση την πρόταση που προβλέπει η Κομισιόν. Το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει σε αυτή την ε, φάση της διαπραγμάτευσης, δηλαδή. Το Συμβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο μπορεί να ορίσει την εντολή διαπραγμάτευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έμπρακτα, αυτό δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να διαβιβάσει τη, τα προσχέδια οδηγιών όχι μόνο στο Συμβούλιο αλλά και στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι απόλυτα λογικό γιατί εφόσον το Κοινοβούλιο έχει τη συνένεση θα πρέπει η Κομισιόν να γνωρίζει ποια είναι τα σημεία που θα ήθελε το Κοινοβούλιο να συμπεριληφθούν στην συμφωνία και εξ αρχής αντί και εξ θα πρέπει να γνωρίζουμε τα δεδομένα. Ιδιαίτερα σε μία διεθνή συμφωνία. Αν και δεν εντάσσεται λοιπόν στη συνθήκη, νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διαβιβάσει τα προσχέδια οδηγιών διαπραγμάτευσης στο Κοινοβούλιο και στις υπεύθυνες επιτροπές που ορίζουν όρους όρους προσυμφωνίας. Αυτό το έκανε η Επιτροπή Ίντε στην έκθεση Λάινεν φέτος το Μάιο για τις επιπτώσεις της συνθήκης της Λισαβόνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτές, αυτοί οι προγενέστεροι όροι σημαίνουν ότι η Επιτροπή θα αντιμετωπίσει την εξή κατάσταση. Θα έχει μία εντολή, μία εντολή από το Συμβούλιο και μία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα θα ήταν σκόπιμο να αποφευχθεί αυτό, να έχουμε μια συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ποιο είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει μια νέα διάταξη που είναι το 218 παράγραφος 10 ότι το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται πλήρως από την Επιτροπή σε οποιαδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων, δηλαδή και εξ αρχής. Και βεβαίως η Επιτροπή πρέπει να το εφαρμόσει αυτό. Δηλαδή σε θέματα εμπορίου τώρα έχουν την ίδια υποχρέωση, δηλαδή να ενημερώνουν το, και το Κοινοβούλιο σε σχέση με την Επιτροπή άρθρου 207 που αντικαθιστά την Επιτροπή του άρθρου 133. Αυτό τι σημαίνει ότι θα ε, υποβλέψουμε το ρόλο της Επιτροπής. Όχι, αυτός δεν είναι ο στόχος. Θέλουμε να ελέγξουμε τι κάνει η Επιτροπή όταν διαπραγματεύεται μία συμφωνία και να ορίσουμε τους βασικούς όρους για το Κοινοβούλιο, αλλά αυτό οπωσδήποτε δεν υποσκάπτει τη θέση της Επιτροπής ως διαπραγματευτή. Δεν είναι αυτό το διακύβευμα, θα πρέπει ίσα ίσα να ενισχύσουμε την θέση της Επιτροπής ως βασικού διαπραγματευτή. Αλλά εάν η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να βρούμε πρακτικούς τρόπους έτσι ώστε εάν το Κοινοβούλιο λάβει πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτή, να μην ε, δημοσιοποιηθούν, διότι αυτό θα είναι εις βάρος των πραγματεύσεων. Για το θέμα του απορρίτου είναι σημαντικό και η Επιτροπή σας θα πρέπει να έρθει σε επαφή με την Κομισιόν έτσι ώστε να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ Κομισιόν και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι δηλαδή οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα δεν θα δημοσιοποιηθούν. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα σε σχέση με το νέο πλαίσιο του δικού σας τομέα. Εάν έχετε αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της ενδεχόμενης συμφωνίας με τις συνθήκες, μπορείτε να ζητήσετε γνωμοδότηση του 10 σε σχέση με την, ε, με την συμβατότητα με τη διαδικασία των συνθήκων, με ό,τι προβλέπουν οι συνθήκες. Το τελευταίο σημείο είναι ένα γενικότερο που αφορά την δυνατότητα που έχουν η ε, ε, Europol, Eurojust και Frontex να συνάψουν διεθνείς συμφωνίες. Αυτό δεν, σημαίνει ότι δεν είναι κατάλληλο, ίσως είναι απόλυτα λογικό και άμεσα αναγκαίο, αλλά θα ήθελα να πω ότι σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις σε σχέση με τη Europol, Eurojust και Frontex, το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει καν, ούτε καν πληροφορείται. Ενώ το Συμβουλίο θα πρέπει να συνενέσει με τη Europol πριν συναυθούν οι διεθνείς συμφωνίες. Αυτό δεν είναι πλέον σύμβατο με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν λέω ότι τώρα θα πρέπει να δράσουμε τάχιστα, αλλά είναι ένα πρόβλημα που ήθελα να θίξω και καθίσατε σαφές ότι χρειαζόσαστε καινούριους κανονισμούς για τη Europol και τη Eurojust, άρα μπορείτε να δείτε το πρόβλημα εκ νέου δηλαδή να θέσετε το Κοινοβούλιο στην, στην ίδια θέση με το Συμβούλιο, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για τις ξεκάθαρες αυτές τις παρατηρήσεις. Να προτείνω το εξής. Προτείνω οι συνάδελφοι να υποβάλουν τα ερωτήματά τους τώρα και τα σχόλιά τους και μετά θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να απαντήσουν εν συντομία. Και μετά θα σας ξαναδώσω το λόγο για να έχετε κι εσείς κάποιο χρόνο να σκεφτείτε τις ερωτήσεις που θα σας τεθούν. Ναι, διαδικαστικό, Κύριε Μπουσουτήλ, ναι, κυρία Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε θα μπορούσαμε να διευκρινίσουμε ότι θα ξεκινήσει η συζήτηση του SWIFT τώρα, γιατί φυσικά αυτά που μόλις μας παρουσιάστηκαν είναι σχετικά με το επόμενο θέμα στην ημερήσια διαταξία, αν σωστά κατάλαβα. Αλλά, όπως είπατε, στην αρχή, στις 10 θα συζητούσαμε το θέμα αυτό. Τι να κάνουμε λοιπόν τώρα, γιατί τα σχόλια τα οποία πολλοί από εμά θα θέλαμε να κάνουμε και οι ερωτήσεις σχετίζονται με τα συγκεκριμένα παραδείγματα της νομικής ερμηνεία, σε ό,τι αφορά την ερμηνεία SWIFT. Τι να κάνουμε λοιπόν κι εμεί. Από μένα εξετάστε λέει η πρόεδρο. Να προτείνω να κάνουμε τον πρώτο γύρο επί των γενικών αρχών, επί των γενικών ε, αν θέλετε συνεπειών. Και νομίζω ότι καλύτερα είναι να συζητήσουμε το SWIFT και τα υπόλοιπα και τις υπόλοιπες συμφωνίες ε, με την παρουσία του, κυρίου Φόλ. Να περιμένουμε στις 10 δηλαδή. Τώρα δηλαδή να ακούσουμε τα πρώτα γενικά σχόλια σε ό,τι αφορά την παρουσίαση που μόλις ακούσαμε, να ακούσουμε και τις απαντήσεις Συμβουλίου και Επιτροπής και μετά μόλις έρθει ο κ. Τζόναθαν Φόλς να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες στις 10. Η Ζανίν Πλάσκατ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο αυτό θέμα, την, ε, το θέμα των ε, οργανώσεων που συνάπτουν διεθνεί συμφωνίε, συμφωνώ ότι δεν ε, συνάδει αυτό με το πνεύμα τη Λισαβόνα και θα θέλαμε να μα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε όντω να αναμένουμε αναθεώρηση των σχετικών κανονισμών. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό και το ανέφερα και χαίρομαι που το αναφέρατε εσείς. Ήταν πολύ σαφής η παρουσίασή σας σαν γέννη. Δεν θα επισέλθω σε θέματα λεπτομεριών σε ό,τι αφορά το SWIFT και το PNR γιατί πρόκειται για συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Αν σωστά όμως κατάλαβε, αν το Κοινοβούλιο δεν συνενέσει η μεταβατική προσωρινή εφαρμογή η οποία προβλέπεται τον Φεβρουάριο εκπίπτει. Θα μπορούσατε να το επιβεβαιώσετε αυτό. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Μπρόγκς είναι επόμενος στον κατάλογο. Ναι, καταρχάς θα ήθελα να ξέρω αν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την ενημέρωση γραπτά. Γιατί... Ναι, την έχετε, την έχετε ήδη στο inbox σας. Σήμερα το πρωί κατέφτασε. Μάλιστα, ωραία. Το δεύτερο ερώτημα. Ακούσαμε ότι αν υπογραφεί μια συμφωνία, φυσικά το Συμβούλιο θα την ολοκληρώσει, θα την συνάψει, εφόσον έχει και την έγκριση του Κοινοβουλίου. Αν δεν έχει την έγκριση του Κοινοβουλίου, τέθηκε το ερώτημα του κατά πόσο το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από το Συμβούλιο να επαναπραδιαγματευτεί. Και νομίζω ότι η απάντηση ήταν αρνητική, γιατί ήδη έχει υπογραφεί η συμφωνία. Είναι αφελής ίσως η ερώτηση, αλλά και τότε τι γίνεται με τη συμφωνία παραμένει έτσι σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Ναι, νομίζω ότι αυτό που ακούσαμε είναι ότι δεν θα τύχει επαναπραδιαπραγματεύσει, αλλά μπορεί να ξεκινήσει νέος γύρος διαπραγματεύσεων, εντελώς νέων. Νέος, ο οποίος φυσικά θα λάβει ε, υπόψη τις προηγούμενες συμφωνίες, μάλιστα. Άρα θα υπερβληθεί. Άρα ουσιαστικά καταργείται. Ναι, ακριβώς, ακριβώς λέει η Πρόεδρος. Αλλά φυσικά θα ληφθεί υπόψη το ότι έχει συμφωνηθεί προηγουμένω. Σάρα Λάτφορντ. Εκτός μικροφώνου. Ναι. Έχασα το πρώτο τμήμα της παρουσίασης, λυπάμαι και ζητώ συγγνώμη. Αλλά νομίζω ότι από αυτά που είπατε θα ήταν θεμητό και επιθυμητό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να έχουν κάπως παρόμοιες απόψεις και δεν είμαι βέβαιη για το πώς θα επιτευχθεί αυτό. Γιατί για συνθήκη μπορούμε να πούμε ότι την δεχόμαστε ή όχι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι α, ας αλλάξουμε αυτό το κομμάτι. Το πρακτικό, αν θέλετε, θετικό στοιχείο είναι ότι δεν έχει η Επιτροπή διπλές οδηγίες. Άρα φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία συνδιαλλαγής. Γιατί δεν είναι άσπρα μαύρα τα πράγματα, δεν είναι απόλυτες οι καταστάσεις. Ποιος μηχανισμός λοιπόν υπάρχει για αυτό την, την, ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Ίσως να μην αναφέρεται ρητά αυτό στη συνθήκη. Θα πρέπει λοιπόν μήπως να τον δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μηχανισμό. Μάλιστα λέει η Πρόεδρος, θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά βλέπω ότι ε, στο ε, έγγραφο που μου δόθηκε περιλαμβάνονται σχετικές οδηγίες. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Θα ήθελα να ενισχύσω και εγώ τις ερωτήσεις που ήδη θέτηκαν σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες, οι οποίες ενδεχομένως θα εμπίπτουν σε αυτή τη μεταβατική φάση μεταξύ Νίκαιας και Λισαβόνας, χωρίς να περάσουμε στο SWIFT. Σε περίπτωση λοιπόν συμφωνιών που έχουν υπογραφεί αλλά δεν έχουν ακόμα συναυθεί, εξ όσων καταλαβαίνω, το Κοινοβούλιο έχει τώρα την αρμοδιότητα να πει ναι ή όχι, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις. Αν θα μπορούσατε να, να μου απαντήσετε σε αυτό, μάλιστα, ο κ. Άλβαρο τελευταίο στον κατάλογο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία μικρή ερώτηση. Με τι πλειοψηφία θα πρέπει να ψηφίσει το Κοινοβούλιο. Απλή, ειδική πλειοψηφία. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό για την όλη διαδικασία. Μάλιστα. Κάνει άλλο συνάδελφο, θέλει το λόγο. Μάλιστα, λοιπόν, να θέσω και εγώ τι ερωτήσει μου οι οποίε απευθύνονται τόσο προ τον κύριο Πάσα από την νομική υπηρεσία αλλά και προ το Συμβούλιο και την Επιτροπή οι οποίοι θα πάρουν το λόγο μετά τη δική μου παρέμβαση. Καταρχάς, μία παρατήρηση. Η πρότασή σας ότι το Συμβούλιο θα πρέπει ανεπίσημα ή σε εθελοντική βάση να διαβουλεύεται με το Κοινοβούλιο για τους όρους τους, ε, της διαπραγματικής νομίζω ότι είναι πολύ λογικό. Γιατί αυτό θα εξασφαλίσει ένα καλύτερο αποτέλεσμα χωρίς ε, να υπάρχουν μετέπειτα αναστατώσεις και αναταραχές Άρα θεωρώ ότι είναι λογικό το αίτημα αυτό και μου είπαν ότι υπάρχει και ο κανόνας 19 του κανονισμού για το πώς θα πρέπει να βρούμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Κατά δεύτερον, και αυτό το απευθύνω κυρίως προς το Συμβούλιο, Μία συμφωνία η οποία βρίσκεται ακόμα σε φάση διαπραγμάτευσης και γίνεται και κλεισμένων των θυρών είναι η άκτα για την παραχάραξη. Και περιλαμβάνονται πολλέ ρήτρε, πολλέ διατάξει, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε, γιατί όλα τα έγγραφα είναι απόρριτα ω συνήθω και κανεί δεν ξέρει, που είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενε. Για παράδειγμα, ρήτρε για την αρμοδιότητα των συνοριοφυλάκων για την ε, κατάσχεση υπολογιστών χωρίς να ακολουθείτε μια ορισμένη διαδικασία. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το Συμβούλιο ποια είναι η αίσθησή του. Μήπως θα μπορούσαν ε, να μας ενημερώνουν σιγά σιγά. Γιατί και εμείς θα πρέπει τελικά να συμφωνήσουμε για αυτές τις διεθνείς συνθήκες σε κάποια φάση. Και να σας παρα πέμψω στο άρθρο 218 σημείο 10 όπου αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάρα αυτά και πλήρως θα πρέπει να ενημερώνεται. Και τέλος, μου άρεσε αυτό που είπατε για τη Europol και τη Eurojust και την ε, Frontex και τη σύναψη διεθνών ε, συμβάσεων. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωκοινοβούλιο απέριψε τέσσερις προτάσεις αναφορικά με τη Europol ως ένδειξη ε, ένστασης. Σχεδόν ομόφωνα. Και μία από αυτές τις συμφωνίες αφορά μια σύναψη διεθνούς ε, συμφωνίας της Europol αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν η χρονική συγκυρία. Και όπως είπα, αυτό θέλω να το σχολιάσει και η νομική υπηρεσία και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω ποιος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπω τον κύριο Μπιάνκι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα είμαι σύντομο από αυτού. Θα ήθελα καταρχά να, να, να ευχαριστήσω τον κύριο Βάσο για την ε, παρουσίασή του, που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και θέτει πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα. Όπω είπαν και πολλοί προηγούμενοι ομιλητέ, η νέα διαδικασία συνένεση σημαίνει ότι, θα να, ότι το Κοινοβούλιο θα μπορεί να πει όχι όταν θα έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Αυτό δεν είναι ο πιο αποτελεσματικό τρόπο κατά πάσα πιθανότητα και νομίζω ότι αυτό που είπαν πολλοί από εσά ότι θα πρέπει να ακούμε τη γνώμη του Κοινοβουλίου εκ των προτέρων είναι ενδιαφέρουσα. Νομίζω θα πρέπει να την εξετάσουμε. Ξέρετε ότι υπάρχει διαθεσμική συμφωνία για το πώς ε, παρέχονται πληροφορίες από την Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Άρα αυτό αποτελεί ένα σημείο εκκίνησης και όπως είπατε και εσείς, Πρόεδρε, υπάρχουν ε, και οι κανονισμοί οι οποίοι έχουν καθιερωθεί για παρόμοιες διαδικασίες σε άλλους τομείς. Νομίζω λοιπόν ότι στην παρούσα φάση δεν μπορώ να επεκταθώ περαιτέρω. Νομίζω ότι πρόκειται για θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν σε διαθεσμικό επίπεδο. Με απότερο στόχο να αποφύγουμε καταστάσεις όπου θα έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και το Κοινοβούλιο θα απαντάει όχι, θα απορρίπτει τις προτάσεις αυτές. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο πλέον αποδοτικός τρόπος. Ευχαριστώ κύριε Μπιάνκη, λέει η Πρόεδρος. Ποιος θα απαντήσει εξ ονόματος του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα θέματα PNR και SWIFT θα τα κοιτάξουμε σε μετέπειτα φάση. Α, δεν θα επισέλθω λοιπόν σε λεπτομέρειες για τα θέματα αυτά από τώρα. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Άκτα, σημειώνω όσα είπατε. Θα τα διαβιβάσω στους συναδέλφους μου. Να δούμε. Μπορεί να σας απαντήσουμε είτε σήμερα αργότερα είτε κάποια άλλη στιγμή. Επιπλέον θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που μόλις ακούστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς έχει η διαδικασία και εμείς ε, ακριβώ έτσι ερμηνεύουμε τη διαδικασία στα πλαίσια του άρθρου 218. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Δεν ξέρω αν ζητά κανεί άλλο το λόγο. Ωραία. Να περάσουμε και πάλι στον κύριο Πάσο. Α, μάλιστα, ζητά ο κύριο Μπρόντ και πάλι το λόγο. Ε, ναι, ναι. Συγγνώμη που λόγο. Μία ερώτηση. νομίζω ότι οι συμφωνίε είναι όλε απόρριτε. Και σε μετέπειτα στάδιο ενημερώνεται το Κοινοβούλιο. Δεν είναι πιο δύσκολο όμως το Κοινοβούλιο να εκφράσει άποψη όταν ξέρει μόνο το γενικό τίτλο και δεν ξέρει λεπτομέρειες. Ναι, ναι, ναι, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι έχετε δίκιο όταν θέτετε το ερώτημα αυτό. Να τη θέσω και εγώ προς την νομική υπηρεσία την ερώτηση αυτή. Φυσικά και θα πρέπει να ενημερωνόμαστε. Δεν είναι δυνατόν να είναι απόρριτα τα θέματα αυτά. Είναι βέβαια επί του παρόντος, αλλά έτσι ανακύπτει το γενικότερο ερώτημα. Τι ποσοστό θα πρέπει να είναι απόρριτο. Γιατί να υπάρχει τέτοιο γενικό κανόνα και να λέει ότι όλε οι διαπραγματεύσει θα πρέπει να είναι απόρριτε. Αυτό φυσικά υπερβαίνει κάπω το πεδίο τη ε, τρέχουσα συζήτηση, αλλά θα το συζητήσουμε. Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ο κύριο Μποζοτήλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το απόρριτο και την ε, Επιτροπή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να ζητήσω από την νομική υπηρεσία να μας απαντήσει για το θέμα αυτό. Έχει την αίσθηση ότι υπάρχει κάποια διαδικασία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα του απόρριτου σε ό,τι αφορά τέτοιες διαδικασίες διαπραγματεύσεων. Υπό το φως φυσικά και του αυξανόμενου ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό και θα θέλαμε να μας πει η νομική υπηρεσία κατά πόσο υπάρχουν ιστορικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση αμα, των εγγράφων και μήπως χρειάζεται αναθεώρηση των διαδικασιών αυτών. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρε. Βλέπω ότι πολλοί ζητούν το λόγο. Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Χένες, να επανέλθω, γιατί ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει Ποιο είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε ό,τι αφορά την σύναψη ε, διεθνών συμβάσεων από διεθνείς οργανισμούς. Δεν μου απάντησε η Επιτροπή, μάλιστα. Να δώσουμε και πάλι το λόγο, λοιπόν, πιο μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Βερζά και μετά ο κύριο Άλμπρεχτ. Ε, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτήν την έννοια της εμπιστευτικότητας. Η συνθήκη της Λισαβόνας ε, δίνει αυξημένες εξουσίες στο Κοινοβούλιο και αν δεν κάνω λάθος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωρίζεται ισότιμα με το Συμβούλιο και την Κομισιόν σε ορισμένους τομείς. Εγώ θεωρώ ότι η έννοια της εμπιστευτικότητας δεν μπορεί να ε, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα έναντι του Κοινοβουλίου κατά τις διαπραγματεύσεις. Ε, να σας πω, ας πούμε, μας έθεσαν ως πρόσχημα την εμπιστευτικότητα για το SWIFT, ενώ ε, το Συμβούλιο τι έκανε, ενημέρωσε τα εθνικά κοινοβούλια τουλάχιστον, αυτό το κάνανε στη Γαλλία και η συμφωνία SWIFT κυκλοφορεί στο ίντερνετ. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα μίνιμουμ ε, σεβασμού που πρέπει να εκφράζεται προς το Κοινοβούλιο και που θα πρέπει να ισχύει. Αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζουμε τα έγγραφα γιατί η Ολλανδική κυβέρνηση δεν ήξερε καν τι είναι το SWIFT και η διαπραγματεύσει ως προς τον εμπιστευτικό χαρακτήρα ε, αυτό είναι ένα ζήτημα. Η διαθεσιμότητα είναι κάτι άλλο, διότι τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες, αλλά θα θέλαμε να γνωστοποιηθούν και στους πολίτες. Η κυρία Ναπολιτάνου ήταν εδώ μαζί μας και ως προς θέμα της ε, εμπιστευτικότητας στην ε, υπόθεση SWIFT εξεπλάγει για το γεγονός ότι το Συμβούλιο αναφέρθηκε στην πλευρά των ΥΠΟ και είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει εμπιστευτικός χαρακτήρας. και άρα το Κοινοβούλιο μπορεί να έχει πρόσβαση στα έγγραφά τους ε, από τη δική του πλευρά. Ο ένας αναφέρεται στον άλλον. ε, τη στιγμή που μιλάμε για έγγραφα τα οποία στα δανείζουν και το Κοινοβούλιο δεν έχει πρόσβαση σε αυτά. Θα πρέπει να πούμε ως Κοινοβούλιο ότι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε επί τέτοιων προτάσεων όταν δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Πρόκειται για μια νομοθετική διαδικασία και θα πρέπει να τη γνωρίζουν τα Κοινοβούλια. Επίσης, αναφερόμενος στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας Δεν ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ελέγχει την εργασία του Συμβουλίου. Αλλά ορισμένα κοινοβούλια πρέπει να έχουν πρόσβαση. Γιατί με ορισμένους φακέλους υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είπα για έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα, το ζήτημα έχει ως εξής. Πολλές φορές τα κοινοτικά θεσμικά όργανα ε, λένε ότι δεν μπορούν να δώσουν έγγραφα διότι υπάρχει συμφωνία εμπιστευτικού χαρακτήρα με τη ΣΥΠΑ. Αυτό έγινε για το PNR αλλά όσα αφορά διαφάνεια και προσπελασιμότητα στα έγγραφα, εμείς είχαμε πληροφορίες από τα, τη ΣΥΠΑ που δεν λάβαμε ούτε καν από το Συμβούλιο, ούτε καν από την Επίτροπη. Θα ήθελα να ρωτήσω απάντηση από το Συμβούλιο ή την Επίτροπη σε σχέση με την Europol και τους άλλους φορείς, την ερώτηση κυρίας Χένες. Το ζήτημα είναι, το ερώτημα το κάλυψα εν μέρη. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Πάσος. Αν αλλάξει η εντολή των γραφείων, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ. No, not very much. In fact, uh, the, the... Δεν έχω κι εγώ να πω πολλά. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς ε, να διευθετήσουμε τα ζητήματα που δεν συζητήθηκαν στο Συμβούλιο. Δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι να ε, δούμε πώς θα διευθετηθεί μελλοντικά. Εάν δεν υπάρχουν άλλα φλέγοντα ζητήματα, θα ήθελα ο κύριος Πάσος να συνοψίσει. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, τέσσερα είδη ερωτήσεων που υποβλήθηκαν. Ε, προσωρινή εφαρμογή, ο ρόλος του Κοινοβουλίου μετά την υπογραφή, το τρίτο, τη συμφωνία ή μη συμφωνία με το Συμβούλιο. Στην πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων, της εντολής και το θέμα ουσίας είναι το θέμα εμπιστευτικό. For the provisional application, the question which was put to be by Mrs. Hennis was what happens with the provisional application if, if that stops now because as we know uh, όπως γνωρίζετε provisional application um... όπως γνωρίζετε ε, και εδώ το βλέπω και στο κατάλογο μου Έχετε 7 συμφωνίες που έχουν υπογραφεί αλλά δεν έχουν συναυθεί. Έχει τον κατάλογο μπροστά σας και το PNR με την Αυστραλία έχει προσωρινή εφαρμογή. Το πρωτόκολλο μεταξύ Ελβετίας, Λίχτενστάιν και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υπογραφεί αλλά έχει προσωρινή εφαρμογή για το κεκτημένο του Σέγγεν το ίδιο ισχύει και για το SWIFT, προσωρινή εφαρμογή και το PNR με τις ΕΠΑ έχει προσωρινή εφαρμογή. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. Εφαρμόζονται λοιπόν οι συμφωνίες με προσωρινή εφαρμογή και θα λήξει μόνο εάν το Κοινοβούλιο πρέπει να συνενέσει ή εάν δεν συνενέσει. Με άλλα λόγια, εάν δεν ε, συμφωνήσει με την ε, συγκεκριμένη συμφωνία και σε αυτήν την περίπτωση η προσωρινή εφαρμογή θα λήξει. Τώρα, ως προς το θέμα που έθεσε ο κύριος Μπουζούτιλ. Ποιος είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου όταν υπογραφούν οι συμφωνίες. Απάντησα διότι δεν μπορείτε πλέον να διαπραγματευτείτε. Έχει γίνει υπογραφή με τρίτες χώρες και το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να πείτε ένα ναι ή ένα όχι. είναι μια πολιτική απόφαση που θα πρέπει να ε, ληφθεί από το Κοινοβούλιο. Βεβαίως είναι πολιτική η απόφαση και δεν θα χρησιμοποιηθεί σε τακτική βάση μέσα στα πλαίσια της ε, υπογραφής ή της προσυπογραφής αυτής. Γι' αυτό θεωρούσα ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερη συνδιαλλαγή με το Συμβούλιο εξ αρχής. Και η βαρόνη Λάντφορτ υπέβαλε το ίδιο ερώτημα. Τι συμφωνία μπορούμε να έχουμε το Συμβούλιο. Θα ήθελα να μιλήσω δυνάμει του 218 που είναι απόλυτα σαφές στην παράγραφο 2 που λέει ότι το Συμβούλιο θα εισαγάγει οδηγίες διαπραγμάτευσης και θα συνάψει συμφωνίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχει τη συνένεση του Συνοβουλίου σε σχέση με τις ε, συμφωνίες αυτές. Άρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις συνθήκες. Αλλά το... αυτό που έχει σημασία είναι και πώς θα τεθούν σε εφαρμογή και πώς μπορούμε να αποφύγουμε μία κατάσταση όπου στο τέλος της διαδικασίας το Κοινοβούλιο δεν θα είναι και ιδιαίτερα ευτυχές με τις διαπραγματεύσεις υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να δεχτεί τη συμφωνία. Αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί εξ αρχής και γι' αυτό είπα ότι τίποτα δεν αποκλεί από την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο, όπως ε, αναφέρεται στο άρθρο 2.18, διότι το προσχέδιο των δύο πραγματεύσεων και το αποστείλει στο Κοινοβούλιο παράλληλα. Και θα υπάρχει έμεση συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την εντολή. Δεν πρόκειται για την διαπραγμάτευση, αλλά για το πλαίσιο. Πώς έχει η εντολή. Τι ζητάμε από την Επιτροπή να κάνει. Διότι η συνένεση είναι το κάτωπτρο της συναπόφασης. Εάν λοιπόν ε, η συνθήκη δεν προβλέπει την συναπόφαση στο πρώτο στάδιο τη εντολής τίποτα δεν αποκλεί από την Επιτροπή να ε, ενημερώσει το Κοινοβούλιο για να γνωρίζει πώς έχει η κατάσταση πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Να γνωρίζει δηλαδή ποιοι είναι οι όροι που θέλει οπωσδήποτε το Κοινοβούλιο. Όπως είπατε, υπάρχει μία ειδική διάταξη, παράγραφος 19 του πλαισίου, που πάει πολύ μακριά, διότι λέει ότι η Επιτροπή διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο το προσχέδιο οδηγιών διαπραγμάτευσης, άρα προτρέχει σε σχέση με, το, με κάτι που ούτε καν τώρα εντάσσεται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Η διάταξη αυτή όμως δεν έχει εφαρμοστεί γενικά για να ικανοποιήσει το Κοινοβούλιο ήδη από σήμερα, από όσο γνωρίζω, διότι όπως ξέρετε στην Επιτροπή Αλίας και στην Ίντε έχετε πολλές ε, διεθνείς συμφωνίες και μας λένε ότι δεν έχουν επαρκείς πληροφορίες. και γι' αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί η όλη πλαισίωση. Τώρα έχουμε μία σαφή διάταξη στην ε, συνθήκη που αναφέρει ότι το Κοινοβούλιο θα πληροφορείται πλήρως σε όλα τα στάδια, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας Νομίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή έχει νομική υποχρέωση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό σε όλα τα στάδια. Τέλος, ως προς το τελευταίο σημείο που είναι ο εμπιστευτικός χαρακτήρας, το άφησα τελευταίο σκόπιμο, σκόπιμα. Γιατί εσείς μιλήσατε ως προς τον εμπιστευτικό χαρακτήρα και είχατε συγκεκριμένη στάση και αυτό ήταν μεγάλη νίκη δική σας η διαφάνεια. Αποτελεί αξία βεβαίως, καμία αμφιβολία, αλλά θα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο για να μην υπονομεύσετε την επιτυχία των διαπραγματεύσεων από την Επιτροπή. Γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να βρείτε μία διευθέτηση, ένα μόντους βιβέντη με την Κομισιόν. Και αυτό το είδα σε σχέση με την ε, με την, το ψήφισμα για την ε, απόρριψη, απέκδηση ευθυνών. Αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει συμφωνία αμοιβαία εμπιστοσύνη έτσι ώστε να δίνουμε πληροφορίες σε όλα τα, τα, θέματα. Και Αυτό που έχει σημασία είναι οι διαδικαστικοί κανόνες για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις, ε, τα, τους φακέλους εμπιστευτικού χαρακτήρα. στο σημείο 3 έχετε το ειδικότερο πλαίσιο το οποίο αφορά μία νέα συμφωνία πλαίσιο που θα πρέπει να τύχει διαπραγμάτευσης και αυτό γίνεται κάθε φορά που αναλαμβάνει την ε, νέα της θητεία η Επιτροπή και αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος της δικής σας επιτροπής δεν χρειάζεται να έχει μία άτυπη συμφωνία με τον υπεύθυνο της Κομισιόν και εδώ σας δίνω το παράδειγμα της Επιτροπής Αλίας και της ΙΝΤΕ διότι προέβησαν σε μία ανταλλαγή επιστολών ή με την ε, Βαρόνη Άστον, με τον κύριο Μπός από την Επιτροπή αλλιές που βελτίωσε την κατάσταση διότι το, διότι δέχτηκε η Επιτροπή να προσέρχεται σε αυτές τις επιτροπές και in camera να δίνει πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Άρα όταν μιλάω για πρακτικές διευθετήσεις, εκεί ακριβώς αναφέρομαι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πάσος. Για θέματα εμπιστευτικότητα συμφωνώ ότι όντω χρειάζεται κάποιο εμπιστευτικό χαρακτήρα για να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Χρειάζεται όμω και διαφάνεια για να υπάρχει εμπιστοσύνη από του πολίτε. Μία τελευταία ερώτηση έχω να κάνω. Αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι σχετίζεται και με την επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε. Το Συμβούλιο όπως λέτε και στις σημειώσεις σας, θα ζητήσει σε εν χρόνο την έγκριση του Κοινοβουλίου, τη συνένεση του Κοινοβουλίου για την σύνεψη διεθνών συμβάσεων. Τι σημαίνει αυτό το εν χρόνο, δηλαδή τι θεωρείτε ότι είναι εύλογη περίοδος, γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει επίσημη προθεσμία και κοιτώντα το PNR, το οποίο προσωρινά ισχύει επί δυόμιση χρόνια, μπορεί να υπάρχει έτσι τέτοια προσωρινή εφαρμογή αόριστα. Υπάρχει κάποιο όριο. Και αυτό το χρησιμοποιώ αν θέλετε και ως σύνδεσμο με την επόμενη συζήτηση γιατί θα είναι πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε πότε μπορούμε να περιμένουμε την επιστολή του Συμβουλίου που θα ζητάει την έγκρισή μας. Πρώτα όμως να μας διευκρινίσετε το νομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το ερώτημα αυτό. Όταν λέω εν ευθέτω χρόνο, χρησιμοποιώ σκόπιμα την έκφραση αυτή, γιατί δεν υπάρχει τέτοια καταληκτική προθεσμία. Δεν υπάρχει χρονικό όριο σε ό,τι αφορά την ε, συνθήκη, αλλά το άρθρο 214 της συνθήκης ορίζει ότι το Συμβούλιο έχει την νομική υπηρεσία, έχει τη νομική υποχρέωση να ζητήσει την έγκριση του Κοινοβουλίου. Αυτό αποτελεί νομική υποχρέωση. Αν υπάρχει λοιπόν νομική υποχρέωση θα πρέπει και να εκτελείται. Το οποίο τι σημαίνει όπως λέτε επειδή κάποιες συμφωνίες ήδη προσωρινά εφαρμόζονται δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να περιμένει ένα χρόνο μέχρι ότου έρθει η επιστολή του Συμβουλίου για να ζητήσει την έγκρισή του λέω τώρα ενδεικτικά ένα χρόνο. Νομίζω ότι το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φυσικά η Επιτροπή θα πρέπει να προετοιμάσει το σχέδιο απόφασης υπό στα πλαίσια του καινούριου άρθρου 218 μπορώ να θέσω και ένα άλλο θέμα το οποίο σχετίζεται με το πρόβλημα μάλλον δεν ξέρουμε αν η Επιτροπή μπορεί να απαντήσει σε τέτοια ερωτήματα στην παρούσα φάση γιατί όπως ξέρετε η Επιτροπή ασχολείται με τις τρέχουσες υποθέσεις. Δεν νομίζω ότι τίθεται όμως τέτοιο θέμα εδώ, γιατί έχουν πλέον ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις. Αυτό που πρέπει να κάνει η Επιτροπή είναι να προετοιμάσει την απόφαση πριν από την σύναψη των συμβάσεων, εφαρμόζοντας αυτά που ήδη υφίσταντο. Δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί νέα πολιτική πρωτοβουλία το οποίο δεν θα μπορούσε να κάνει η Επιτροπή υπό τις παρούσες συνθήκες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος. Νομίζω ότι αυτά ήταν χρήσιμα και εν ώψη της ε, επόμενης συζήτησης. Ελπίζω να μπορέσετε να μείνετε για να απαντήσετε τις ερωτήσεις οι οποίες ενδεχομένως να ανακύψουν από την επόμενη συζήτηση και να καλωσορίσω τον κύριο Τζόναθαν Φόλα από την Επιτροπή και τον κύριο Χένιγκαρ εκ μέρους της Σουηδικής Προεδρίας. Αν θα θέλετε να κάνετε μια σύντομη εισαγωγή, γιατί ανακοινώθηκε στην ατζέντα ότι το θέμα αυτό αφορά μόνο το SWIFT, αλλά τα ίδια θέματα ανακύπτουν και σε διαφορά αφορά το PNR. Αν θα θέλετε να πείτε και κάτι για το άκτα, παρακαλώ, γιατί τις ίδιες ερωτήσεις θα θέσουμε και για το άκτα. Και αν θα μπορούσατε επίσης να απαντήσετε κάποια ερωτήματα που τέθηκαν για το τελευταίο ζήτημα, το πότε μπορεί να περιμένουμε δηλαδή την επιστολή αίτησης έγκρισης. Και να δώσω το λόγο στον κύριο Φόλ πρώτα. Ευχαριστώ, καλημέρα σας και σας εύχομαι μια καλή Λισαβόνα. Δεύτερη ημέρα λοιπόν, σήμερα. Δεν έχουμε ακόμα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Χαιρόμαστε όμως ιδιαίτερα που πλέον υπάρχουν ερωτήσεις που καλούμαστε να απαντήσουμε. Εδώ στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να δώσουν, αν θέλετε, νόημα στη νέα μας συνθήκη. Ασφαλώς η Επιτροπή είναι δεσμευμένη σε ό,τι αφορά την στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, προκειμένου από κοινού να αναπτύξουμε στον τομέα της ΚΕΠΑ τον χώρο ασφάλισης και δικαιοσύνης που μας απασχολεί. Αυτό φυσικά, όπως ξέρετε, περιλαμβάνει και πολλές διεθνείς αλλά και εγχώριες ε, εσωτερικές διαδικασίες. Είναι η δεύτερη ημέρα λοιπόν της Λισαβόνας και είναι ασφαλώς και μία ιδιαίτερη ευαίσθητη χρονική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί όπω είπε και ο συνάδελφο από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε μια φάση υπηρεσιακή αν θέλετε. Σύντομα θα μάθουμε ποιοι είναι οι δύο επίτροποι για τη Δικαιοσύνη και τις ιστορικέ Υποθέσεις και θα πρέπει να είναι προσεκτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς οι υπάλληλοι ιδιαίτερα για να μην, ε, αν θέλετε, προδικάσουμε το τι θα θελήσει να κάνει η καινούργια επιτροπή. Τι θα θελήσουν να έρθουν να σας πούν οι καινούργιοι επίτροποι. Αλλά φυσικά δεν ε, ενεργούμε και σε κενό αέρος, δεν είμαστε αφελείς. Ξέρουμε ότι έχουν ήδη πάρει το δρόμα τους διάφορες ενέργειες, διάφορα προγράμματα και ότι όντως πριν από κάποιες ημέρες το Συμβούλιο έλαβε σημαντικές αποφάσεις τις τελευταίες ημέρες της ισχύω της συνθήκης της Νίκαιας και οι συνέπειες αυτών των αποφάσεων θα συζητηθούν σήμερα. Η Επιτροπή θα υιοθετήσει σήμερα την επανομαζόμενη ανακοίνωση Omnibus που θα περιλαμβάνει λεπτομερώς όλες τις πράξεις που εκκρεμούν μετά την Δευτέρα το βράδυ και θα εξηγήσει σε εσά και στο Συμβούλιο ποιες είναι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιες θα είναι δηλαδή οι νέες προτάσεις, οι οποίες δεν θα ακολουθήσουν φυσικά πάρα αυτά, αλλά τέλος πάντων θα δρομολογηθούν ποιες προτάσεις εκκρεμούν μετά τη λήξη της συνθήκης της νίκαιας. Και θα τα ανακοινώσουμε αυτά στο Κοινοβούλιο με την κανονική διαδικασία. Οι πιο πολλές εκκρεμούσες προτάσεις θα αντικατασταθούν από καινούργιες, στο σύντομο δυνατό. Και λυπάμαι που χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις που δεν είναι πολύ ωφέλιμες, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα θα, πότε θα αναλάβει καθήκοντά της Νέα Επιτροπή. Δεν ξέρουμε λοιπόν πότε θα βγούμε από αυτή την ενδιάμεση κατάσταση της υπηρεσιακής, αν θέλετε, Επιτροπής. Ελπίζουμε σύντομα στις αρχές του επόμενου έτους. Ωστόσο, ασχολούμαστε και δουλεύουμε εντατικά στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Σε επίπεδο λοιπόν υπηρεσιών, προτιμάζουμε, προκειμένου να προτείνουμε στους νέους επιτρόπους να υποβάλουν πολύ γρήγορα προτάσεις, διαδικασίες, για παράδειγμα σε ποινικά ζητήματα, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, της εκμετάλλευσης των παιδιών, για παράδειγμα. Όλα αυτά αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες και δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι δεν θα παραμείνουν κορυφαίες προτεραιότητες. Αυτά λοιπόν θα πράξουμε και πριν ολοκληρώσω θα ήθελα να σχολιάσω και λίγο από τη συζήτηση την οποία είχα την τιμή να ακούσω πριν από λίγο. Ασφαλώς και θα υποβάλουμε προτάσεις προς το Συμβούλιο, προκειμένου το Συμβούλιο να ζητά την έγκριση του Κοινοβουλίου για διεθνείς συμβάσεις. Αυτό θα το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν και αυτό και πάλι εξαρτάται από το πότε θα ξεκινήσει, θα αναλάβει τα καθήκοντα της η νέα Επιτροπή αυτό εξαρτάται και από πολλές πρακτικές πτυχές, όπως για παράδειγμα τη μετάφραση των κειμένων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος όμως να καθυστερούμε την εφαρμογή των συμφωνιών αυτών και θέλουμε να γίνει η εφαρμογή αυτή με την πλήρη δημοκρατική έγκριση του Κοινοβουλίου. Προετοιμάζουμε λοιπόν τις διαδικασίες αυτές προκειμένου να μπορέσετε το συντομότερο δυνατόν να συμβάλλετε σε αυτή την δημοκρατική διαδικασία. Δεν μπορώ όμως να δεσμευτώ για το χρονικό πλαίσιο, να είστε όμως βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ουδεμία επιθυμία να καθυστερήσει τη διαδικασία και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και τη συμφωνία SWIFT θα ισχύσει ούτως ή άλλως μόνο για εννέα μήνες. Άρα, λίγαν συντόμως θα επανέλθουμε στο Συμβούλιο με πρόταση για να μας δοθεί διαπραγματευτική εντολή για τη σύναψη νέα συμφωνίας και το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει με το φυσιολογικό τρόπο που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας και μας ανέφερε η νομική υπηρεσία τι προβλέπει το κείμενο της νέας συνθήκης. Λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τέτοιες διεθνείς διαπραγματεύσεις. Θα έχουμε λοιπόν ευκαιρίες για να θέσουμε αυτή την ε, νέα πορεία την οποία μόλις τώρα ξεκινάμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Να καλέσω, να δώσω το λόγο στον κύριο Χένιγκερ από το Συμβούλιο για να μας διαφωτίσει για τις μελλοντικέ μας συνεργασίες, να μας πει ιδιαίτερα πότε μπορούμε να αναμένουμε την επιστολή που θα ζητήσει την έγκρισή μας. Θα ξεκινήσετε να μας ενημερώνετε κατευθείαν για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για το ΑΚΤΑ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές. Θα ήθελα καταρχάς να πω σε ό,τι αφορά το φάκελο του SWIFT εκτιμήσαμε ιδιαίτερα τη στενή συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών σε ό,τι αφορά Είχαμε έρθει πολλές φορές εδώ στην Επιτροπή και ακούσαμε πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από εσάς σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τον Ιούλιο και ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα είμαι σύντομος. Δεν θα ήθελα άλλωστε να επαναλάβω τα όσα μας είπε ο Τζόναθαν Φόλ από την Επιτροπή. Είναι λοιπόν η πρώτη ημέρα της Συνθήκης Λισαβόνας. Είναι ακόμα λίγο νωρίς λοιπόν να απαντήσουμε λεπτομερώς τις ερωτήσεις σας για το πότε θα λάβετε τις σχετικές πληροφορίες. Ωστόσο, να σας ενημερώσω ότι η Προεδρία δεν σκοπεύει σε καμία περίπτωση να καθυστερήσει τη μεταφορά της προσωρινής συμφωνίας, τη διαβίβαση της προσωρινής συμφωνίας προς το Κοινοβούλιο για την έγκρισή της θα πρέπει φυσικά να ολοκληρώσουμε και να πάρουν την οριστική της μορφή τα αποτελέσματα, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η συζήτηση στα πλαίσια της Επιτροπής του άρθρου 36 για την μεταφορά, τη διαβίβαση του κειμένου αυτού. Στην Επιτροπή ΚΑΤΣ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε και ο Τζόναθαν Φόλ. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί αναφορικά με τους ρόλους, αναφορικά με το πώς και πότε θα διαβιβαστεί η απόφαση αυτή στο Κοινοβούλιο. Ασφαλώς το συντομότερο δυνατόν. Πρόεδρε. Πρόεδρε, θέσατε και το ερώτημα του ΑΚΤΑ. Απάντησα και προηγουμένως ότι δεν είμαστε σε θέση εδώ και τώρα να εκφραστούμε ή τουλάχιστον εγώ δεν είμαι σε θέση να εκφραστώ εδώ και τώρα λεπτομερώς να τοποθετηθώ για το άκτα. Ίσως ε, μια καλή ευκαιρία να ήταν στις 7 Δεκεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα κατά τις διαβουλεύσεις. Θα σταματήσω λοιπόν στο σημείο αυτό και ασφαλώς είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Μάλιστα, ευχαριστώ. Βλέπω ότι ήδη πολλοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Μία διευκρίνηση μόνο. Είπατε ότι το Συμβούλιο θα συζητήσει την επόμενη εβδομάδα τον τρόπο και τη διαδικασία που θα ζητήσει την έγκριση του Κοινοβουλίου. Αυτό αναφέρεται και στο SWIFT και στο PNR. Ναι, σε κάθε περίπτωση έχει να κάνει με τη συμφωνία SWIFT και φυσικά στο σχετικό πλαίσιο τίποτα δεν μας εμποδίζει να συζητήσουμε και για τη συμφωνία PNR. Αλλά βασικά το βασικό θέμα είναι, θα είναι η συμφωνία SWIFT. Okay, do... Μάλιστα, αλλά υποθέτω ότι το ίδιο θα γίνει και για το PNR ή μάλιστα να το θέσω αλλιώς, μάλλον να το θέσω αλλιώς, να συστήσω να γίνει αυτό και το, για το PNR. Ο κύριος Άλβαρος ζήτησε πρώτα στο λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ, ευχαριστώ γιατί και το Συμβούλιο μας ε, έδωσε απαντήσεις. Τώρα για να συνοψίσω από ό,τι κατανοήσαμε θα πρέπει να συνενέσουμε. Δεν ξέρω όμως ποιος θα μας δείσει η συνένεση, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή. Α, το Συμβούλιο, το Συμβούλιο. Γιατί αναρωτιέμαι ως προς το χρονοδιάγραμμα ότι, και φαντάζομαι ότι ε, δεν θα είναι δύσκολο, διότι το 218 λεει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συμφωνήσουν σε ένα χρονοδιάγραμμα συνένεσης. Άρα θα πρέπει να ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Και σε περίπτωση απόρριψης, ας πούμε, από το Κοινοβούλιο, πώς θα ε, στραφούμε προς τις νέες ε, διαπραγματεύσεις. Δηλαδή θα έχουμε ε, συναπόφαση με συμμετοχή του Κοινοβουλίου ή μέσα στα πλαίσια μίας ε, διεθνούς συμφωνίας. Θα διαπραγματευτούμε με τις ΣΥΠΑ και μετά θα ζητήσουμε τη συνένεση του Κοινοβουλίου. Γιατί σε αντίθεση με την Επιτροπή Αλίας αυτό δεν το κάνουμε και πολύ συχνά. Το θέμα του άκτα θα ήθελα μία εκτίμηση από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή σε σχέση με αυτά που μας είπαν και είναι φήμες, γιατί κανένας δεν είδε τη συμφωνία. Θα έχουμε ένα σύστημα ηχνηλασιμότητας σε παγκόσμιο ε, επίπεδο, αλλά αυτό είχε ε, απορριφθεί τέσσερις φορές και στις τηλεπικοινωνίες το διαγράψαμε οριστικά. Δεν θα ήταν ε, παραβίαση του κοινοτικού κεκτημένου εάν σε παγκόσμιο επίπεδο ε, το εντάξουμε αυτό σε μια συμφωνία και θα μας ε, πλήξει διότι στην ουσία αντιτασσόμεθα στο νομικό μας πλαίσιο. Έχω ορισμένα ονόματα, αλλά έχασα και μερικούς. Mr. Busuttil, Mr. Albrecht, anybody else asked for the floor? Ludford? And it's Mr. Um, Okay, I would, I would like to ask you to, to all... Θα ήθελα όλοι σας να μην υπερβείτε τα τρία λεπτά. Η κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία ερώτηση την οποία έθεσε και ο κύριος Άλβαρο. Ακούσαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί από το Συμβούλιο και θα τους ζητηθεί η έγκριση από το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά το SWIFT, αλλά από ό,τι ακούσαμε η Επιτροπή θα συστήσει στο Συμβούλιο να το κάνει αυτό. Ρωτώ λοιπόν, μπορεί το Συμβούλιο από μόνο του να ζητήσει την έγκρισή μας ή χρειάζεται σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί τότε τίθεται το ερώτημα το κατά πόσο μπορεί να το κάνει αυτό η υπηρεσιακή ε, επιτροπή ή θα πρέπει να περιμένουμε την καινούργια επιτροπή. Μιλήσαμε σήμερα για το SWIFT αλλά δεν θα ήθελα να ξεκινήσω επί του περιεχομένου συζήτηση για τη συμφωνία SWIFT αλλά εκφράσαμε τις ανησυχίες μας και τις αμφιβολίες μας και είπαμε ότι το Κοινοβούλιο σήμερα μόνο ναι ή όχι μπορεί να πει και μας είπαν ότι είναι το σύστημα γκυλοτίνα. Θεωρώ ότι αυτό για το Κοινοβούλιο αποτελεί μια κατάσταση η οποία είναι διόλου ικανοποιητική, η οποία τονίζω όμως θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, γιατί ξέρουμε εδώ και καιρό ότι αυτό το μήνα θα τεθεί σε ισχύ η Λισαβόνα. Άρα με λίγη καλή θέληση και με καλή, με λίγη εμπιστοσύνη μεταξύ των επιτροπών θα μπορούσαν ε, να έχουμε θα μπορούσε να έχει συμμετάσχει πιο πολύ το Κοινοβούλιο τους τελευταίους μήνες της εργασίας και θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε αποφύγει να τεθεί σε, να υπογραφεί λίγες ώρες πριν την θέση σε ισχύ της Συνθήκης Λισαβόνας ή η συμφωνία αυτή Κατά το παρελθόν, σε πολλές περιπτώσεις ε, ακούγαμε τον όρο εμπιστευτικές ε, διαπραγματεύσεις και τώρα έχουμε το εξής πρόβλημα. Πώς θα διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες, πώς θα τις συζητήσουμε του καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα και ελπίζω όντως στο μέλλον να διαμορφωθούμε με διαφορετικό τρόπο αυτές οι συζητήσεις, αυτές οι διαδικασίες. Ευχαριστώ, κυρία Χένες. Θα ήθελα να μιλήσω περισσότερο στο περιεχόμενο της συμφωνίας SWIFT. Θα ήθελα ο Τζόναθαν Φόλ να με διαφωτίσει στο θέμα της αμοιβαιότητας, διότι προσπάθησα να κατανοήσω την αρχή της, αμμο... της εμπιστοσύνης, αλλά δίνουμε πρόσβαση στα δεδομένα στις ΕΠΑ Ζητάμε από τις υπηρεσίες των ΙΠΑ να μας δώσουν πληροφορίες Όπως είπα και σε προγενέστερες συζητήσεις, εμείς δεν έχουμε το δικό μας TFTP ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι η αρχή της αμοιβαιότητας δεν υπάρχει. Αυτό το επιβεβαίωσαν ορισμένα κράτη-μέλη. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε θέματα αμοιβαιότητας. Σε σχέση λοιπόν με το θέμα του συστήματος οικονομικού εντοπισμού τρομοκρατών και το θέμα της αμοιβαιότητας, αυτό που έχει σημασία είναι και το ψήφισμα που εγκρίναμε ε, το Σεπτέμβριο. Τι, γιατί μιλάμε τώρα αρμόδια αρχή, δικαιοδοτική αρχή και τι ε, εντολή έχει οι αρμοδιότητες. Αλλά στο προσχέδιο ελέγχθη ότι εάν ο ε, πάροχος δεν μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τεχνικούς λόγους, όλα τα στοιχεία θα ε, μεταφερθούν στην αρμόδια αρχή, θα μεταφερθούν συλλήβδιν στη δημόσια αρχή. Ε, ο κύριος Μπουζούτιλ. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ στη δήλωση της Προεδρίας σε σχέση με τη στενή συνεργασία που είχε με το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει όμως να σας πω ότι δεν εκτιμώ το γεγονός ο, για το πώς έχει χειριστεί το θέμα η Προεδρία με την απόφαση που ελήφθη την προηγούμενη Δευτέρα. Αναφέρομαι στην επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου στις 26 Νοεμβρίου ε, ζητώντας ρητά από την Προεδρία να διαγράψει αυτό το σημείο από το Συμβούλιο Υπουργών αυτή τη βδομάδα. Και αυτό διότι όλοι γνωρίζαμε ότι η νέα συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ και συνεπώς Θέλαμε μια θετική ανταπόκριση από το Συμβούλιο για να διαβιβάσει το μήνυμα ότι για το Συμβούλιο η νέα συνθήκη αποτελεί ε, πολιτική διαφοροποίηση καθώς και μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας. Αντί για αυτό, η απάντηση που έλαβε ο κύριος Μπούζεκ δύο μέρες ε, μετά ήταν ε, η απόρριψη του αιτήματό του. Άρα θα ήθελα μια ε, διασαφήνιση της θέσης του Συμβουλίου επί του θέματος και επίσης θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα θα πρέπει να μεταφερθεί σε υψηλότερα επίπεδα από αυτήν την Επιτροπή γιατί έχει γίνει ένα διαθεσμικό ζήτημα όπου έχουμε τον πρόεδρο της δικής μας Επιτροπής, ε, το αίτημα το οποίο ε, απερίφθη από το Συμβούλιο την ίδια ημέρα θέσει σε ισχύ στη συνθήκη, δηλαδή λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η νέα συνθήκη. Άρα το Συμβούλιο αγνοεί το, το Κοινοβούλιο και τώρα μας λέει να έτσι έχουν τα πράγματα. Είτε το δεχόσαστε είτε το απορρίπτετε. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό το στάδιο. Εάν αυτό είναι ένα προμήνυμα των μελλοντικών καταστάσεων, εμείς θα πρέπει να ε, δείξουμε, να επιδείξουμε τη δική μας ευθύνη και να χρησιμοποιήσουμε τις ε, αρμοδιότητες ε, δυνάμεις της συνθήκης, της συνθήκης και δεν θα αποτραβηχτούμε από αυτό. Πέρα από το περιεχόμενο της συμφωνίας, αλλά αυτό είναι θέμα κάθε αυτό που ορίζει, που οδηγεί σε σημαντικά προβλήματα σε σχέση με τη διαθεσμική συνεργασία και θα ήθελα ε, μια διασάφηση επί του περιεχομένου. Και εδώ θα ήθελα πάλι να το ζητήσω αυτό από την νομική υπηρεσία η οποία α, παρίσταται. Θαύμα. Καταρχήν, ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας, θα πρέπει να εκτιμήσουμε πώς ε, θα ληφθεί υπόψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια αυτής της ε, ε, συμφωνίας. Και αυτό θα πρέπει να το αναλύσουμε πριν φτάσουμε στο ζήτημα για το κατά πόσο θα αποφανθούμε καταφατικά ή αρνητικά. Θα πρέπει όμως να είμαστε σίγουροι να γνωρίζουμε κατά πόσο έχουν ανταποκριθεί στα αιτήματά μας. Ως νομική υπηρεσία θα ήθελα να πω τι θα γίνει αν απαντήσουμε αρνητικά. Ποιες θα είναι οι συνέπειες ως προς τη, την εφαρμογή της ε, προσωρινής συμφωνίας και ποια προστασία για τους πολίτες θα εφαρμοστεί εάν η προσωρινή εφαρμογή δεν ισχύει πλέον. Αυτό με απασχολεί ιδιαίτερα στην ε, περίπτωση που θα αποφανθούμε αρνητικά, διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε τις συνέπειες οποιασδήποτε ενδεχόμενης ε, αποφασής μας. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω κατά πόσο η Βελγική Συμφωνία θα εφαρμοστεί και πώς θα επηρεάσει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις συναλλαγές SWIFT. Και θα ήθελα να ρωτήσω λήψη οποιασδήποτε συμφωνίας μαζί και της προσωρινής, τι επίπεδο προστασίας διαθέτουν οι πολίτες επί του θέματος. Άρα κύριε Μπουζουτήλ μας λέτε ότι επειδή εμείς χειριζόμαστε την ε, γιλιοτίνα, ίσως το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να μας σκοτίζει και ιδιαίτερα. Άλμπρεχτ. Δεν χαίρομαι. Να συνεργάζομαι με την Προεδρία του Συμβουλίου στο με το SWIFT και άλλους διότι με ανησύχησε αυτό που συνέβη τη Δευτέρα και σε άλλους τομείς όπως το Europol διότι είχαμε τέσσερις αποφάσεις από το Συμβούλιο με συμφωνία 90% από όλες τις ομάδες και δεν λάβαμε απάντηση δηλαδή το Συμβούλιο ενέκρινε το ολοπλαίσιο. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι ο σωστός ε, τρόπος διεκπεραίωσης της εργασίας και επειδή μιλάμε και για εμπιστοσύνη στον ε, τομέα του απορρίτου, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στην εργασία του Συμβουλίου και καμία διαφάνεια. Δεν μπορώ να εμπιστεύομαι το Συμβούλιο ούτε καν στις διαπραγματεύσεις ε, σύναψης συμφωνιών. Και αυτό είναι πρόβλημα για μας, διότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης όπου κάπου που να μπορούμε να πούμε ωραία σε αυτό το πλαίσιο ως κοινοβούλιο ε, αναθέτουμε μία εντολή και στην περίπτωση της άκτα δεν λειτουργεί έτσι η δημοκρατία Όπως ε, γνωρίζουμε τώρα, υπάρχει κάτι σαν την άκτα. Α, και λέει το Συμβούλιο, ωραία, ελάτε τώρα να το συζητήσουμε. Πρέπει να συμμετέχουμε στην όλη διαδικασία και όπως, είπε, η, όπως αναφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας, στο μέλλον θα πρέπει να είμαστε πλήρως εμπλεκόμενοι. Αυτό σημαίνει στην περίπτωση SWIFT ότι υπάρχουν πολλά τμήματα όπως τα παραρτήματα για το τι περιλαμβάνεται για τα στοιχεία SWIFT-FIN, κατά πόσο περιλαμβάνονται γιατί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δεδομένων ίσως εμπλέκονται περισσότεροι φορείς και χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να το απορρίψει. Bronze. Εκτός ε, μικροφώνου. Άμε συγχωρείτε. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ και σε προγενέστερες συζητήσεις, αλλά ως προς το θέμα της συμφιλίωσης του θέματος ε, εμπιστευτικού χαρακτήρα και αμοιβαιότητας, ε, πιστεύω ότι το αρχικό κείμενο θα πρέπει να ε, διαβάσετε στο Κοινοβούλιο, αλλά το περιεχόμενο μετέπειτα, συ, ε, μετέπειτα διαπραγματεύσεων παραμένει εμπιστευτικό. Δηλαδή, θα γνωρίσουμε ποιο είναι το θέμα, τουλάχιστον αυτό. Ένα ερώτημα που υποβάλλατε στη νομική υπηρεσία εσείς αφορούσε το μέλλον των ρητρών αυτοεξαίρεσης της Δανίας, Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου από τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Από ό,τι άκουσα, η νομική υπηρεσία δεν μπορεί να αποφανθεί. Δεν ξέρω κατά πόσο οι εκπρόσωποι της Σουηδικής Προεδρίας και του, της Κομισιόν μπορούν να σχολιάσουν. Η κυρία Βέρζε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα ξεκινώντας με... Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα διαδικαστικό. Λοιπόν, τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας και είμαστε αρκετοί εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο που ήμασταν εναντίον της συνθήκης και αναρωτιέμαι αλλά πόσο καιρό θα θριαμβολογούμε πια πολλοί βουλευτές καταψήφισαν εθνικοί και ευρωβουλευτές την ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά η κοινή γνώμη επίσης καταδίκασε σε μεγάλο βαθμό. Πόσο καιρό λοιπόν θα θριαμβολογείται. Εγώ, ξέρετε, ήμουνα υπάλληλο, δημόσιο υπάλληλο στη χώρα μου και θεωρώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να εκφράζουν μία σχετική εγκράτεια, δεν θα πρέπει να συγκρατούνται, δεν μπορούν να εκφράζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι τόσο ελεύθερα τη γνώμη τους θριαμβολογώντα. Στην ομάδα μου πια έχουμε βαρεθεί αυτές τις ε, θριαμβολογίες. Οι περισσότεροι από εσάς θριαμβολογείται γιατί αυξάνονται οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι και εγώ γιατί ποτέ μου δεν πολέμησα αυτήν την πλευρά της συνθήκης. Αλλά θεωρώ ότι τα πράγματα εξελίσσονται πολύ άσχημα εδώ. Ε, για, ως προς την ε, με, μελλοντική μεθοδολογία εργασίας εγώ θεωρώ ότι αυτή η τρικέφαλη εξουσία που προδιαγράφεται θα πρέπει να κερδίσει κατά πολύ σε δημοκρατικότητα αν θα πρέπει, αν θέλουμε μάλλον να γίνει αρεστή από τους ε, πολίτες. Για το SWIFT Το Κοινοβούλιο τόνισε πάντοτε το θέμα της προστασίας των πολιτών και οι επιφυλάξεις που εκφράσαμε είναι οι μικρές δυνατότητες, οι ανισότητες ε, δυνατότητας προσφυγής ε, των πολιτών. όταν ε, βρίσκονται στην Αμερική ή στην Ευρώπη. Ο επόπτης που πρότειναν άλλοι συνάδελφοι δεν βοηθάει σε τίποτα. Εγώ πιστεύω απλώς ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την προστασία των δεδομένων των πολιτών. Και για αυτά που είπαν ο κύριος Μπουσουτήλ και ο κύριος Άλμπρεχτ. Δεν θα έπρεπε να διαμαρτυρηθούμε για την περιφρόνηση που εξέφρασε το Συμβούλιο της προάλλες και έναντι της SWIFT και έναντι της Ευρωπόλ. Εμείς στείλαμε ένα μήνυμα προς το Συμβούλιο και για το SWIFT και για την Ευρωπόλ. Αλλά μας αγνώρισαν παταγωδός. Και αυτό κάνουν συστηματικά. Μάλιστα ενδυναμώνουν και τη θεωρία της συνωμοσία. Δεν θα πρέπει εμείς να θεσπίσουμε τέτοιου είδους σχέσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος θριαμβολογίας. Έχετε δίκιο. Αλλά όλοι θεωρούμε ότι είναι ένα βήμα προς τα μπρος για την ε, διαφάνεια και τη δημοκρατία και την ε, επιρροή του, του πολίτη ως προς θέση σε ισχύ της Συνθήκης Λισαβόνας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η Επιτροπή τους τελευταίους μήνες είδε τους τελευταίους μήνες πώς ε, πρέπει να κινηθούμε στο επόμενο επίπεδο. Αυτό το καλωσορίζουμε όλοι και ξέρω ότι και, εσείς το κάνετε. Ο κύριος Βος. Ευχαριστώ. Καταρχάς, ε, βλέπω τους εκπροσώπους των δύο άλλων θεσμικών οργάνων, δεν τους βλέπω καθόλου να θρέμβολογούν. Βλέπουμε, λοιπόν, ε, και αναρωτιόμαστε τι έγινε, δεν ξέραμε δηλαδή 30 30-12 επρόκειτο, επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή η πρώτη δεκάτου της Σύνδικης της Λισαβόνας. Ε, Εμείς ευθυνόμαστε που δεν είχαμε ενημερωθεί. Γιατί στην τελική ανάλυση ήταν, ε, προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι η Τσεχία υπέγραψε στην τελική ανάλυση τη συνθήκη της Λισαβόνας και τελικά ε, βρεθήκαμε σε μια κατάσταση την οποία δεν μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει. Θα ήθελα όμως να λάβετε υπόψη τη νέα κατάσταση η οποία ισχύει από χτες και να μην ξεχνάμε διάφορες τρέχουσες καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να μας απασχολήσουν και στην επόμενη διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα διαθεσμικά όργανα. Και ίσως αυτό θα ήταν και μια εργασία για την ε, διαθεσμική συμφωνία, μια αμοιβαία υποχρέωση ενημέρωσης σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από αυτό το συναισθηματικό, αν θέλετε, και θεσμικό στοιχείο, θα ήθελα να διαχωρίσω τα στοιχεία επί του περιεχομένου και θα ήθελα να σας διασφαλίσω ότι η απόφασή μου για το ναι ή όχι, την έγκριση ή μη έγκριση, δεν θα επηρεαστεί από την ε, διαθεσμική αυτή πτυχή. Άλλο πράγμα η διαδικασία και άλλο το ποια θα είναι η συνέπεια αν απορρίψουμε την πρόταση. Και νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή οι πολίτες θα βρεθούν σε μια νομική κατάσταση η οποία θα είναι χειρότερη από το περιεχόμενο το οποίο προς το παρόν ακόμα δεν το γνωρίζουμε αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μια πρώτη δήλωση για το πώς θα συνεχιστεί, πώς θα διεκπαιρεωθεί η κατάσταση και τι θα γίνει αν απορριφθεί αυτή η πρόταση και πώς έχει η νομική κατάσταση σε περίπτωση τέτοιες απόρριψης για τον πολίτη. Για το κατά πόσο θα υπάρξει στην Ευρώπη ένα τέτοιο σύστημα TFTP ή ε, κατά πόσο δεν θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα ήταν αρκετά σημαντικά για να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και το θέμα του πώς διασφαλίζεται ότι οι εμπειρίες που έλαβαν οι αρχές των ΙΠΑ και οι γνώσεις που έχουν για σχετικά ζητήματα αν θα διαβιβαστούν προς εμάς για να μπορέσουμε και εμείς έτσι να αντιδράσουμε. Uh, Ευχαριστώ κύριε Φως. Θεωρώ ότι αν η συμφωνία SWIFT απορριφθεί δεν υπάρχει συμφωνία, άρα δεν υπάρχει συμφωνία για τη μεταφορά δεδομένων. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Κύριε Σταβάρη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας, θίγοντας ένα θέμα διαδικαστικό, πολιτικό, αλλά και περιεχομένο. Για τους εννέα μήνες που ακούμε συνεχώς. Φαίνεται ότι αποτελεί αυτό ένα από τα πιο αδιάσυστα στοιχεία της ε, Επιτροπής του Συμβουλίου, ότι πρόκειται τους ή άλλους για προσωρινή συμφωνία, θα ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μετά από εννέα μήνες. Τι θα συμβεί όμως στα στοιχεία που θα έχουν ήδη συλλεχθεί κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών, γιατί η συμφωνία προβλέπει την τήρηση, την κράτηση των στοιχείων επί πέντε έτη, υποκωδικοποιημένη και κρυπτογραφημένη μορφή σε περίπτωση που χρειαστούν τα στοιχεία αυτά μετά από, για παράδειγμα, τρομοκρατική επίθεση. Τι θα γίνει λοιπόν με τα στοιχεία αυτά που θα συλλεχθούν. Θα κρυθούν επί πέντε έτη. Δηλαδή τι, ρισκάρουμε να κρατηθούν τέτοια στοιχεία με τη μέχρι όσο ανακύψει μια κυβέρνηση τύπου Σαρα Πέιλιν. Πάντα είναι πιο εύκολο να φυλάμε τέτοια στοιχεία παρά να κάνουμε ένα διαχωρισμό, μια διαγραφή κάποιων εξ αυτών. Άρα αυτό το διαδικαστικό θέμα συμπεριλαμβάνει και ένα θέμα επί της ουσίας. Εμπιστευόμαστε τις αρχές. Εμπιστευόμαστε να τηρήσουν οι αρχές επί πέντε έτη τα στοιχεία αυτά. Επίσης, δεν πρόκειται να ξαναξεκινήσουμε μετά από εννέα μήνες από την αρχή γιατί τα θεσμικά όργανα θα έχουν ήδη θέσει κάποιες πρακτικές τις οποίες θα έχουν συνηθίσει πιο απλό θα είναι να κρατήσουμε μετά από εννέα μήνες τις ίδιες πρακτικές θα υπάρχει ήδη μία συμφωνία η οποία θα αποτελεί τη βάση μίας μετέπειτα συμφωνίας χωρίς καμία αμφιβολία και θα βρεθούμε σε φάση αναδιαπραγμάτευσης με την Αμερικανική κυβέρνηση για μια συμφωνία η οποία ήδη υφίσταται. Άρα, είμαι μεν αισιόδοξο, αλλά δεν θεωρώ ότι αν ακολουθήσει νέα συμφωνία βάσει της προσωρινής συμφωνίας θα μπορέσουμε να αλλάξουμε πιο πολλά. Θα αλλάξουμε μόνο λεπτομέρειες. Και αυτό που με ενοχλεί ιδιαίτερα είναι ότι το Κοινοβούλιο έχει προειδοποιήσει επαντελημένα τις άλλες ε, πλευρές, τα άλλα μέρη, ότι θέλουμε να ακολουθήσει η διαδικασία αυτή τη συνθήκη της Λισαβόνας, ακόμα και αν δεν είχε ακόμα εφαρμοστεί η Λισαβόνα. Εδώ και καιρό είχαμε απευθύνει τις, τις προειδοποιήσεις αυτές, άρα πώς μας κατηγορείτε ότι αντιδρούμε με τον τρόπο της γκυλοτίνας. Τίφονται πρακτικά θεσμικά και διαδικαστικά ζητήματα. Η Τζανίν μίλησε για αμοιβαιότητα από τη ΣΥΠΑ. Γιατί ξέρουμε πάντα όταν διαπραγματευόμαστε συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ ότι υπάρχει ο κίνδυνος να απορριφθεί η συμφωνία αυτή από το Κογκρέσο και αυτό το λαμβάνουν όλοι υπόψη στη φάση διαπραγμάτευση συμφωνιών με τις ΗΠΑ. Μήπω ήρθε ο καιρό να το έχουμε αυτό υπόψη μα και σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρε, Μιλάμε για την κοιλωτίνα, αλλά έχουμε καταργήσει την θανατική ποινή στην Ευρώπη. Αυτό είμαι σίγουρη ότι καθησυχάζει την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Έχουν ζητήσει οι συνάδελφοι να ταυτερολογήσουν, αλλά έχουμε ήδη καθυστερήσει. Δεν είναι πρόβλημα φυσικά αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση, αλλά σας παρακαλώ δεν θέλω να ακούσω ε, δηλώσεις, θέλω να ακούσω ερωτήσεις. Μάλιστα, ένα λεπτό. Το ξέχασα προηγουμένω, ο κύριος Άλβαρο. Πότε θα λάβουμε αυτό το έγγραφο για την ε, έγκρισή μας. Θα λάβουμε το πλήρες έγγραφο προς έγκριση ή υπάρχουν μήπως ε, κρυφά παραρτήματα για το SWIFT για παράδειγμα. Θα λάβουμε και τα απόρριτα συσσαγωγικά έγγραφα, γιατί φυσικά θα πρέπει να αποφασίσουμε επί του συνόλου του πακέτου. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε επιμερών αυτού. Η κυρία Σίπολ. Ευχαριστώ. Μία μικρή παρατήρηση πριν κάνω την ερώτησή μου. Να σταματήσει πια αυτή η συζήτηση στο Κοινοβούλιο που έχουμε θέσει πολλές φορές ε, ασφάλεια των πολιτών έναντι προστασία των πολιτών. Σας παρακαλώ, μία ερώτηση λέει η Πρόεδρος. Γι' αυτό λοιπόν να κάνω και την ερώτησή μου. Τι θα συμβεί αν το Κοινοβούλιο πει όχι. Έχει ελέγξει κανείς από το Κοινοβούλιο, από την νομική υπηρεσία, από την Επιτροπή σε περίπτωση τρομοκρατικών επιθέσεων θα υπάρχει σχετική προστασία, ανάλογη προστασία και υπάρχει κάποια απόδειξη ότι η συμφωνία αυτή και τη η διαδικασία την οποία επί 8 έτη εφαρμόζουν οι ΙΠΑ είναι όντως ε, σωστή και αποτελεσματική. Ευχαριστώ συνάδελφος, λέει η Πρόεδρος, για τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει, ποιος θα ήθελε να πάρει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πάλι πολλές ερωτήσεις υποβλήθηκαν και θα προσπαθήσω να ασχοληθώ με τις περισσότερες. Και όπου παραλείψω κάτι θα με πλαισιώσει η Επιτροπή. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι και έτσι κατανόησα και εγώ την παρέμβαση της νομικής υπηρεσίας δεν θα υπήρχε διαφορά ως προς την επιρροή του Κοινοβουλίου με το κατά πόσο αυτή η συμφωνία έχει υπογραφεί τις 30 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου, οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία. Όπως και να έχουν τα πράγματα, θα πρέπει να συνενέσει το Κοινοβούλιο ή να απορρίψει. Και υπ' αυτή την έννοια Οι επιστολές που έχουν αποσταλεί και εδώ αναφέρομαι στην επιστολή του κυρίου Μπούσεκ προς τον Πρωθυπουργό μου και την απάντηση της Σουηδικής Προεδρίας και ως προς την νομική κατάσταση η οποία σκιαγραφήθηκε σε αυτή την επιστολή ε, Κοινοβούλιο δεν στερείται των δικαιωμάτων του, όπως αναφέρθηκε στην επιστολή Μπούζεκ. Και επίσης για τη μακροχρόνια συμφωνία, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνενέσει ενδεχομένως. Η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό μου και προς την Προεδρία καθορίζει την αξία και τη σημασία του προγράμματος από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι κάτι που αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι η εντολή εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο καθώς και η Συμφωνία. Τώρα έχουμε ένα άλλο καθεστώς λήψης αποφάσεων δυνάμει της συνθήκης ε, της μας. ομόφωνα Ομόφωνα αυτό σημαίνει και τα τέσσερα κράτη-μέλη που απήχαν. Ναι, ναι, ναι. Η ομοφωνία ε, σημαίνει ή ότι ψηφίζει κανείς καταφατικά ή ότι απέχει. Αυτό σημαίνει αμόφωνη απόφαση. Ως προς το περιεχόμενο, αυτή η συμφωνία, μάλλον το TFTP ισχύει από το 2001 και επαναλαμβάνω το πρόγραμμα του Συστήματος Εντοπισμού Τρομοκρατών ισχύει από το 2001 και ε, δεν υπάρχει αλλαγή ως προς την εμβέλεια της συμφωνίας. Δεν πρόκειται για περισσότερα στοιχεία, διαφορετικά στοιχεία. Έγινε λόγος για τα στοιχεία ΣΕΠΑ, τα οποία ποτέ δεν απεστάλησαν, ούτε χρησιμοποιήθηκαν. Αλλά και ούτε και αποκλείονται. Τα μηνύματα ΦΙΝ ε, υπάρχουν. Εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονος σε, σε συναλλαγές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ισχύει λοιπόν αυτή η προσωρινή συμφωνία που θα έχει τις ε, ίδιες, ε, του, την ίδια εμβέλεια στο μέλλον. Ως προς την προστασία δεδομένων έχει επέλθει βελτίωση ως προς τις ρήτρες διασφάλειας, ε, θέματα αμοιβαιότητας, θέματα αποκατάστασης. Ίσως η Σουηδική Προεδρία θα έπρεπε να έχει διαπραγματευτεί καλύτερα. Δεν είχαμε τόσο ε, καλή κάλυψη της αμοιβαιότητας αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια βελτίωση σε σχέση με την προγενέστερη κατάσταση. Γι' αυτό συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι η συμφωνία αυτή βελτιώνει την κατάσταση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό ήταν και ο απότερος στόχος μας. Ανέκαθεν. Ως προς ε, ένα TFTP της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συστήματος εντοπισμού τρομοκρατών δηλαδή. Αυτό δεν ε, επίκειται, αλλά άκουσα να λέγεται από το κοινοβόλιο θα πρέπει να υπάρχει ένα TFTP σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ένα σύστημα οικονομικού εντοπισμού τρομοκρατών. Ως προς θέματα εμπιστοσύνης και εμπιστευτικού χαρακτήρα, απλώς επαναλαμβάνω ε, το ότι τα απόρριτα έγγραφα θα τα βλέπουμε με το Κοινοβούλιο και αυτό έχει ε, σχέση με θέματα εμπιστοσύνης. Ως προς την άκτα, κύριε Άλβαρο, Είπατε ότι κανένας δεν έχει δει το κείμενο. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω για το φάκελο άκτα σήμερα. Ε, οι διαπραγματευτές και δεν ξέρω κατά πόσο υπήρξε διαρροή του φακέλου. Ε, είναι λυπηρό αυτό, αλλά αυτό ισχύει πολλές φορές. Κύριε Άλμπρεχτ, μιλήσατε για τη Europol και για το SWIFT. Το Συμβούλιο έλαβε αποφάσεις εφαρμογής Αυτές οι αποφάσεις ε, εφαρμογής ε, αποφασίστηκαν ως σημείο α στο Συμβούλιο στα πλαίσια της Europol από πρώτης πρώτη, πρώτου. Χωρίς αυτές τις αποφάσεις θα είχαμε βασικά ελλείμματα στη λειτουργία της Europol από την 1η Ιανουαρίου. Ως ε, Προεδρία κατανοήσαμε από το Συμβούλιο ότι είναι πολύ σημαντικός αυτός ο φορέας. Γι' αυτό προωθήσαμε τις ε, συναφείς συμφωνίες. Βεβαίως ε, η κατάσταση έχει αλλάξει άρδιν σήμερα. Η Europol διέπεται από μία σύμβαση Είναι κάτι λοιπόν ότι είναι, αυτό αποτελεί βελτίωση για το μέλλον. Ξέρω ότι δεν απάντησα όλες τις ερωτήσεις και πιστεύω ότι ο Τζόναθαν Φολ θα σας ε, καλύψει περισσότερα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ που ήσασταν τόσο πλήρης και σε διαφορά γύρω. τη Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε που, για το ότι είναι σημαντικά τα θέματα αυτά και γι' αυτό είναι σημαντικό να ενημερώνεται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Θα αλλάξει όμως η διαδικασία στο μέλλον. Κύριε Φόλου. Um, ευχαριστώ. Πριν απαντήσω στις ερωτήσεις, να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή για την υπόθεση αυτή. Γιατί μπορεί να έχουμε ξεχάσει πως στάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Αυτό το σύστημα λειτουργούσε με μυστικό τρόπο για κάποια χρόνια. Ναι, δεν είμαι βέβαιος ότι το ξέρουν όλο αυτό, όλοι αυτό. Δεν υπήρχε καμία προστασία δεδομένων. Υπήρχε απόλυτη μυστικότητα. Εκτός από μία συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και μετά από αίτηση του Βέλγου Πρωθυπουργού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε να εξετάζει το θέμα αυτό και τώρα βάσει εντολής του Συμβουλίου και κατά συμμόρφωση με αποφάσεις ε, του Κοινοβουλίου της 17 Σεπτεμβρίου έχουμε συνάψει μια συμφωνία με όποιες ατέλειες ε, έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχουν η Προεδρία και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει ένα λίγο διαφορετικό αποτέλεσμα. Καταφέραμε ωστόσο να πετύχουμε μια συμφωνία την οποία με προθυμία θα προτείνουμε στο Συμβούλιο να ζητήσει την έγκριση του Κοινοβουλίου. Ο, τζατ, ο δικαστής Μπριγκέρ έχει παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα μιας λεπτομερούς ανάλυσης για το τι συνέβη. Αν θέλετε, θα να μιλήσω και κλείσμο ένα των θυρών, προτείνω να μιλήσετε με τους ειδικού, με τους εμπειρογνώμονες για τα θέματα τα τρομοκρατικά των κρατών μελών σας. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν τέτοιες υπηρεσίες και αυτοί για τη δική μας ασφάλεια και την ασφάλεια όλων μας χρησιμοποιούν τα στοιχεία του TFT. Αυτό είναι λοιπόν το σημείο κίνηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, είναι χρήσιμο, λειτουργεί και γι' αυτό προτείνουμε να συνεχιστεί. Ποτέ δεν αποκρύψαμε από το Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία μέχρι το τέλη του έτου λόγω της απόφασης του SWIFT να μεταβιβάσει, να μεταφέρει τα δεδομένα. Κανεί δεν σχεδίασε να γίνει αυτό πριν από την θέση σε ισχύ της Λισαβόνας για να εξαπατήσουμε το Δεκέμβριο. Και το Σεπτέμβριο προσπαθήσαμε να το εξηγήσουμε αυτό. Θέλατε να υπάρχει περιορισμός μέχρι 12 μηνών. Θέλατε να υπάρχει και διαμόρφωση στα πλαίσια της Λισαβόνας. Και αυτό ακριβώς σας δώσαμε και μάλιστα όχι 12 αλλά 9 μήνες, 3 μήνες λιγότερους. Άρα μην σκεφτείτε ούτε κατά διάνοια ότι κάποιος σκόπιμα ή έστω από αμέλεια ήθελε να εξαπατήσει το κοινοβούλιο αυτό. Δρούμε υποπλήρη διαφάνεια διαφάνεια. το δεύτερον, τι θα συμβεί αν ε, δεν δώσετε την έγκρισή σα. Θα το δούμε αυτό, αλλά προφανώ η συμφωνία δεν θα τεθεί σε ισχύ. Και ποιο θα πληχθεί. Εγώ θεωρώ, με όλο το σεβασμό, η ασφάλεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πληχθεί και η προστασία των δεδομένων, γιατί φαντάζομαι ότι οι Αμερικανοί θα βρουν τρόπους να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία για τους Ευρωπαίους που θέλουν, χωρίς καμία δικλίδα ασφαλείας. Πόσο θα διαρκέσει δεν ξέρω, γιατί υπάρξει νέα συμφωνία πολύ σύντομα. Ίσως καλύτερη συμφωνία, ίσως με καλύτερες διαπραγματευτές και θα είναι υπεύθυνοι η Κομισιόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε καλύτεροι στη διαπραγμάτευση από τη Σουδική Προεδρία. Θα υπάρξει λοιπόν νέα συμφωνία μετά από έγκριση του Κοινοβουλίου. Αλλά έχει δίκιο ο Πρόεδρος. Ε, Γκυλοτίνα ημί. Αυτός είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου για τις διεθνείς συμβάσεις είναι να τις συγκρίνει ή να μην τις συγκρίνει. Είναι κάπως δεσμευτικό. Αλλά έτσι γίνεται. Δεν διαπραγματεύονται τα κοινοβούλια τις συνθήκες αυτές. Σε τελική ανάλυση το κοινοβούλιο θα εγκρίνει ή δεν θα εγκρίνει τη συμφωνία. Έτσι είναι χωρισμένες οι νομοθετικές εξουσίες. Αλλά σε τελική ανάλυση θα δώσετε την έγκρισή σας ή δεν θα τη δώσετε. Πρόκειται για μια σημαντική εξουσία, για μια σημαντική ευθύνη. Για την αμοιβαιότητα. Δεν έχουμε TFTP στα κρατημέλη μας. Και εξ όσων γνωρίζω, κανείς δεν είναι διτεθειμένος να δαπανίσει τα υψηλά κονδύλια που χρειάζονται για να δημιουργήσει ένα τέτοιο σύστημα. Δεν ξέρω αν θα δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό TFTP, σύστημα οικονομικού εντοπισμού τρομοκρατών. Γιατί αλλάζουν ε, και οι επίτροποι, αλλάζει και ο πρόεδρος και το καθεξής. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ περίπλοκο ακριβό σύστημα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό ότι χρησιμοποιούμε δωρεάν το αμερικανικό σύστημα για να σας μιλήσω με πάσα ειλικρίνεια σε ένα βαθμό ναι. Λαμβάνουμε τέτοια στοιχεία από τη ΣΥΠΑ, οι οποίες μεταξύ άλλων στοιχεία τα οποία τη χάνουν με το σύστημα SWIFT. Και θα σας πούν όλοι ότι είναι χρήσιμα αυτά τα στοιχεία σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας. Άρα θα έπρεπε να πω και να παραδεχτώ ότι υπάρχει μια ασύμετρη αμοιβαιότητα, γιατί δεν έχουμε σύστημα PNR. Προτείνουμε ένα σύστημα, όχι πάρα πολύ γρήγορα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε κάτι τέτοιο ακόμα. Οι Αμερικανοί έχουν τέτοιο σύστημα και μας παρέχουν κάποιες πληροφορίες. Μιλάμε για μια περιορισμένη λοιπόν αμοιβαιότητα η οποία συνάδει και πάλι με την εντολή που μας έδωσε το Συμβούλιο. Με ρωτήσατε για την ε, διάταξη αναφορικά με την προμήθεια δεδομένων Συλλήβδιν. Ξέρετε νομίζω πώς λειτουργεί το σύστημα, το SWIFT. Δεν γνωρίζει τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που κάνουν συγκεκριμένες συναλλαγές ούτε σε πρώτη φάση το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν ούτε το TFTP λόγω των συστημάτων προστασίας δεδομένων που προβλέπονται για το σύστημα αυτό. Άρα τι συμβαίνει. Στη ΣΥΠΑ ζητείτε προμήθεια ζητείται να παραχθούν, να χορηγηθούν ένα σύνολο πληροφοριών. Πάντα για τις ανάγκες συγκεκριμένης έρευνας. Και μετά εξετάζεται το σύνολο αυτό των πληροφοριών και αναζητούνται ενδεχομένως λεπτομέρειες που μπορεί να είναι και προσωπικά δεδομένα. Μόνο όμως αν τα άτομα αυτά συνδέονται με μία συγκεκριμένη έρευνα. Γι' αυτό μιλάμε για συλλήβη, παροχή στοιχείων. Άρα, οι πιο πολλοί από εμά είμαστε ένας αριθμός. Και τα προσωπικά μας δεδομένα, η ταυτότητά μας δεν μπορεί να εξακριβωθεί, αλλά είναι κάπως ηρωνικό, ακριβώς επειδή υπάρχει προστασία των δεδομένων, έτσι δουλεύει το σύστημα αποκαλύπτουμε μόνο έγγραφα στο Κοινοβούλιο. Α, συγγνώμη, αν θα αποκαλύψουμε έγγραφα στο Κοινοβούλιο, ε, ναι, το χρόνο, ναι, πότε ακριβώς δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι διαθεσμικό ε, ζήτημα υψηλού επίπεδου. Πώς θα συμβεί τώρα ακριβώς αυτό? Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε και σίγουρα όταν θα πρέπει να ζητήσουμε την έγκρισή σας θα σας υποβάλουμε όλα τα στοιχεία, όλα τα έγγραφα για τα οποία θα συζητήσουμε την έγκρισή σας. Για το συγκεκριμένο ερώτημα του τι συμβαίνει με τα δεδομένα τα οποία ήδη θα έχουν συλλεχθεί όταν θα ανασταλεί ή τερματιστεί η συμφωνία. Αυτό προβλέπεται συγκεκριμένα στο 14.2 της συμφωνίας. Σε περίπτωση ακύρωσης, ε, κατάργησης ε, των, της συμφωνίας, όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την Αμερικανική κυβέρνηση θα τύχουν ε, επεξεργασία μεταχείρισης σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας. Αυτό περιλαμβάνει και την προστασία των δεδομένων. Ακόμα και σε περίπτωση που θα καταπέσει η συμφωνία αυτή. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν θα υπόκεινται στους στην εφαρμογή των όρων αυτών, συμπεριλαμβανομένη τη διαγραφή των στοιχείων αυτών. Γι' αυτό που ρώτησε η κυρία Ζίπελ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε, αν θέλετε, αντάλλαγμα που μπορούμε να κάνουμε μεταξύ πολιτικών ελευθεριών και προστασία. Εμεί στην Επιτροπή και η μελλοντική μου Επίτροπη που θα είναι υπεύθυνη για τον τομέα αυτό, ξέρω ότι υπάρχουν γενικά και αόριστα δηλώσεις για την ισορροπία μεταξύ των δύο στοιχείων, αλλά αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να εκπληρώσουμε και τις δύο α, συνιστώσεις της πολιτικής. Να προσφέρουμε την ασφάλεια που προαπαιτείται με τον παράλληλο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θεωρούμε ότι αυτό το έχουμε πράξει και το ίδιο έκρινε ομόφωνα και το Συμβούλιο. Και όντως η αποχή αποτελεί ε, μέθοδο ομόφωνης συνένεσης. Το κατά πόσο λειτουργεί ή δεν λειτουργεί τώρα η συμφωνία. Σας παρακαλώ να λάβετε στα σοβαρά την απόφαση του δικαστή Μπρουσιέρ, γιατί όντως έχει αποφασιστεί, έχει εξακριβωθεί ότι υπάρχει πολιτικό όφελος και αν δεν την ακολουθήσουμε θα έχουμε σπαταλήσει πολύ πολιτικό κόπο. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, ορισμένα ζητήματα που παραμένουν. Ε, το ένα ερώτημα του κυρίου Μπουζούτη λόγω προς συμφωνία με το Βέλγιο και η δική μου ερώτηση προς την Επιτροπή υποθέτω για το κατά πόσο το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις ΑΚΤΑ. Και θα ήθελα να πω ότι αν η συμφωνία SWIFT απορριφθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί ή ε, άλλα κράτη δεν έχουν ε, πρόσβαση στην πληροφόρηση, απλώς θα είναι πιο περίπλοκο, πιο ε, βαρύ το σύστημα. Μπορείτε να απαντήσετε κύριε Φόλ, μπορείτε να απαντήσετε και στις δύο για την άκτα. <coughs> Δεν έχω λεπτομεριακή ε, πληροφόρηση. Δεν ξέρω κατά πόσο ο βοηθός μου μπορεί να συνδράμει εδώ. Όχι, δεν αφορά τη δική μου γενική διεύθυνση. Μετά από την ε, ολοκλήρωση της ε, συμφωνίας θα ενημερωθείτε πλήρως. Αλλά ο συνάδελφος από τη Γενική Γραμματεία θα σας μια απάντηση από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Λυπάμαι λοιπόν. Δεν περίμενα μία τέτοια ε, ερώτηση. Λοιπόν, Βέλγιο, Βέλγιο. Και ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές. Η ε, αρμόδια αρχή είναι το δικαστικό σύστημα του Βελγίου, το οποίο, από το οποίο θα ζητηθεί αμοιβαία αρρωγή από τη ΣΥΠΑ και θα την αντιμετωπίσουμε κατά τον συνήθι τρόπο. Εδώ θα πρέπει να προσέξω τα λόγια μου, όπως είναι γνωστό. Γιατί επιλέγουμε το Βέλγιο, γιατί το SWIFT εντοπίζεται στο Βέλγιο, αλλά η βάση δεδομένων που περιλαμβάνει οι συναλλαγές SWIFT που θα αποτελέσουν αντικείμενο μεταφοράς η βάση δεδομένων ε, βρίσκεται σε ένα άλλο κρατός μέλος που δεν απέχει χίλια χιλιόμετρα από το Βέλγιο αλλά αυτό το κράτος λέει ότι πρέπει να αναφέρουμε το όνομά του. Ε, τότε μην το αναφέρετε. Ε, πολύ ωραία χώρα είναι βέβαια. Υπάρχουν ε, συμφωνίες και διευθετήσεις μεταξύ των δύο χωρών έτσι ώστε τα στοιχεία που ζητάμε από ένα βελγικό δικαστήριο αυτά τα στοιχεία θα αποσταλούν στο Βέλγιο γι' αυτό τον ε, λόγο. Αυτή η χώρα που δεν αναφέρεται, ε, αυτή τη χώρα την οποία δεν αναφέρεται, τη γνωρίζω πολύ καλά, το ίδιο και η κυρία Χένες. Αυτό που έχει σημασία είναι το γεγονός ότι η χώρα αυτή δεν είχε καμία σχέση με το θέμα, αλλά υπάρχει κακή επικοινωνία. Έχουμε καθυστερήσει. Θα μπορούσε η νομική υπηρεσία να επανέλθει εν συντομία και να μας απαντήσει ο κύριος ε, Πάσος. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Πάσος. Σε σχέση με το, τα παράπονα του κυρίου Μπουζούτιλ που είναι απόλυτα κατανοητά γιατί εάν δεν υπεγράφει η συμφωνία την 30 ε, ε, Νοεμβρίου, το Κοινοβούλιο θα βρίσκεται σε μια διαφορετική θέση και ίσως σε, συμμετέχει πιο ενεργά στις διαπραγματεύσεις ή τουλάχιστον ενημερώνεται καλύτερα. Τώρα που έχουν λήξει οι διαπραγματεύσεις, έχω ένα ερώτημα. Δεν κατανόησα όπως είπε ο Τζόναθαν Φόλο, τι θα συμβεί με τη συμφωνία SWIFT εάν λάβουμε υπόψη και το ανακοινωθέν τύπου από το Συμβούλιο, διότι αυτή η συμφωνία που υπογράφει την 30 Νοεμβρίου θα ισχύσει προσωρινά από την 1η Φεβρουαρίου 2010 και θα λήξει στις 31 ε, Οκτωβρίου 2010 εκτός και εάν χρησιμοποιήσετε το άρθρο 14 της Συμφωνίας για ρήτρα αναστολής. Δεν ξέρω κατά πόσο το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνενέσει σε αυτή τη συμφωνία και αν ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Συμβούλιο. Διότι ο κύριος Φόλ μας είπε ότι η Επιτροπή ήδη το Φεβρουάριο προετοιμάζει μία σύσταση για την επόμενη συμφωνία, δηλαδή τη μακροχρόνια συμφωνία. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έχει η κατάσταση για αυτή τη συμφωνία και θα πρέπει να το γνωρίζει το Κοινοβούλιο και αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ο Τζόναθαν Φόλο να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Γνωρίζουμε όλοι εδώ ότι η συνθήκη της Λισαβόνας υπεγράφει δύο χρόνια πριν. Άρα δεν με εκπλήσει να ακούω από το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να δούμε τρόπους εφαρμογής για να δούμε πώς το Συμβούλιο θα ζητήσει τη συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά πρέπει να προετοιμαζόμαστε συνεχώς και όχι να αρχίσουμε την επόμενη εβδομάδα με την Επιτροπή 36. Αυτό το λέω γιατί όπως υπενθύμησε ο κύριος ε, Πάσος, η συμφωνία SWIFT θα τεθεί σε ισχύ το Φεβρουάριο και από νομικής πλευράς δεν υπάρχει κανένα πρόσκομα έτσι ώστε να αποσταλεί η συμφωνία της 30 Νοεμβρίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει κανένα πρόσκομα έναντι αυτού. Αυτή είναι υποχρέωση. Δεν πρόκειται για θέμα αμοιβέ εμπιστοσύνη. Το άρθρο 218 αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε επίγουσες καταστάσεις μπορούν να συμφωνήσουν ως προς το χρονικό περιορισμό και πιστεύω ε, ότι δεν υπάρχουν νομικά προσκόμματα για να μην αποστείλουμε ήδη πριν από την 1η Φεβρουαρίου, εν πάση περιπτώσει, ε, ένα αίτημα συνένεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι συμφωνούμε απόλυτα ως προς το θέμα εμπιστευτικού χαρακτήρα, διότι έχουμε μία διμερή διαθεσμική συμφωνία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε σχέση με θέματα απορρίτου. Άρα έχουμε όλα τα μέσα έτσι ώστε να λαμβάνουμε ε, έγγραφα απόλυτα εμπιστευτικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη διασάφηση και ήταν χρήσιμη γιατί αυτό θα ήθελα να πω και εγώ Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει, αλλά δεν έχουμε και πολλά στην ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση ως προς τη μεταβατική περίοδο. Δηλαδή, η 1η Δεκεμβρίου δεν ήταν και έκπληξη. Γι' αυτό θα περίμενα από το Συμβούλιο ως υπεύθυνο όργανο να μας έχει ήδη προετοιμάσει αυτό το αίτημα συνένεσης με βάση το νομικό υπόβαθρο που μόλις μας σκιαγράφησε η Νομική Επιτροπή. Θα μπορούσατε να απαντήσετε εντάχει σε αυτό το ερώτημα και να μας εγγυηθείτε ότι θα λάβουμε ένα τέτοιο αίτημα το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Όπως ήδη είπα, ο Τζόναθαν Φόλ συμφώνησε μαζί μου Αυτό το θέμα θα αποσταλεί στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια συζήτηση για, τον ε, τρόπο, για τους τρόπους αποστολής και αυτή η διαδικασία συνένεσης θα αναλυφθεί από το Κοινοβούλιο. Αυτό θα γίνει ταχύστα. Σας είπα ότι προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε την Επιτροπή καθεαυτή, καθώς και τα μεμονωμένα μέλη της Επιτροπής. Και υπήρξε μια πρόσκληση σε γεύμα, την οποία επαναλαμβάνω έτσι ώστε να το δούμε το θέμα στο υπόλοιπο της Προεδρίας μας. Τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε γραπτός διότι δεν είναι άκρος ικανοποιητικά. Δεν νομίζω ότι η άτυπη πληροφόρηση one-to-one ε, είναι πλήρως ενημερωτική. Εάν θα πρέπει να αποφασίσουμε για κάτι, θέλουμε πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα επί των οποίων ε, αποφασίζουμε. Και προτείνω να ζητήσουμε αίτηση συνένεσης επί όλων των διαδικασιών. Φολ. Θα ήθελα να κατανοήσετε κάτι. Ε, φαίνεται σαν να μπήκαν όλα στη θέση τους ε, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα της 30 Νοεμβρίου. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν ήμασταν σίγουροι ότι είχαμε ε, ε, συμφωνήσει με τις ΗΠΑ. Και όπως ξέρετε, δεν ήταν σίγουρο το Συμβούλιο θα συμφωνούσε. Θα κάνουμε δύο πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το κάνει το Συμβούλιο, αλλά εμεί θεωρούμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει ε, την ε, απόδοση, μάλλον την ε, επιζήτηση συμφωνίας. διότι θα κρατήσει για εννέα μήνες στην περίπτωση που θα συνενέσετε. και θα το κάνουμε αυτό. Και το Συμβούλιο θα σας δώσει όλες τις ε, πληροφορίες έτσι ώστε να ακολουθήσετε τις δύο διαφορετικές διαδικασίες. Με βάση την 30 Νοεμβρίου και παράλληλα Θα γνωρίζετε τη διαδικασία του Συμβουλίου έτσι ώστε να έχετε πώς έχουν τα πράγματα και ο διαπραγματευτής θα σας κρατήσει ενημέρωση για το 218 10 με βάση τις διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, ένα τελευταίο, μία τελευταία ερώτηση. Είπατε στην αρχή της παρέμβασής σας ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να το κάνει αυτό τη στιγμή που είναι μια ενδιάμεση επιτροπή, υπηρεσιακή επιτροπή. Δεν μπορώ να σας δώσω μία τελική απάντηση, διότι όλα εξαρτώνται από τις ε, νομικές συμβουλές που αναμένουμε από τη νομική υπηρεσία, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή ως υπηρεσιακή Επιτροπή. Άρα, ίσως αυτό είναι θέμα για την επόμενη Επιτροπή, αλλά αυτό απέχει μόνο λίγες εβδομάδες εγώ θα έλεγα δύο μήνες λέει η πρόεδρος, τέλος πάντων. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να εγκρίνει ή να λάβει απόφαση το συντομότερο δυνατόν και ελπίζω η Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεωρήσουν ότι πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία που μας απασχολεί εδώ και μήνες και είναι δυνατόν να λάβουμε μία απόφαση υπό την τρέχουσα επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Α, θα παραμείνετε και στο επόμενο, για το επόμενο σημείο. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, έχουμε δύο ακόμα θέματα που απομένουν στην ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Πόλη θα κάνει μια σύντομη εισαγωγή για τα δύο θέματα αυτά. για το 19 και το 20, τα τελευταία δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ, αν φύγετε από την αίθουσα, κάντε ησυχία. Okay. Uh, colleagues, shall we first and briefly deal with the, the question because Mr. Fall Συνάδελφοι, να κοιτάξουμε πρώτα το θέμα αυτό. Γιατί ο κύριος Φόλ μπορεί να απαντήσει το θέμα που θέσαμε και χτες για τον προπολογισμό και την ε, Επιτροπή του Άρθρου 39. Επίσης, να μας πείτε πώς επηρεάζει η συνθήκη της Λισαβόνας την δικαστική συνεργασία και την αστυνομική συνεργασία καθώς και τα δικαστικά θέματα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα για το πρώτο θέμα, για το άρθρο για την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 που έχει δημιουργηθεί από τις Διευθύνσεις για την Προστασία Δεδομένων. Προβλέπει ότι το άρθρο 29 της Επιτροπής θα πρέπει να παρέχει γραμματιακή υποστήριξη στις υπηρεσίες, γιατί η ομάδα δεν έχει προϋπολογισμό. Δεν έχει προπολογισμό και η Επιτροπή, όπως πολύ καλά ξέρετε, δεν μπορεί να δημιουργήσει σχετικούς προϋπολογισμούς. Είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνει μια μεγάλη αναθεώρηση και συζήτηση για τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ελπίζω να τροποποιήσουμε σημαντικά την οδηγία για το άρθρο 29 που πλέον έχει, είναι πολύ παλιά και τώρα από ο τρίτος πυλώνας έχει μειωθεί κατά μεγάλο βαθμό. Να σκεφτούμε τουλάχιστον να υπάρχει ένα ενιαίο μέσο για την πλευρά την εμπορική αλλά και την αστυνομική δικαστική της προστασίας των ε, προσωπικών δεδομένων. Και φυσικά θα ξανασυζητήσουμε τον σκοπό και τη λειτουργία της ομάδας Επιτροπής, της Επιτροπής ε, ε, ε, του άρθρου 29, αλλά δεν είναι συμβουλευτική επιτροπή. Δεν αποτελεί, δεν υποκαθιστά τον Ευρωπαίο επόπτη για τα, ευρωπαϊκά, για τα προσωπικά δεδομένα. Έχει συγκεκριμένο ρόλο, τον οποίο και δεν πρέπει να υπερβεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα το οποίο σχολίασα και κατά την εισαγωγή μου Ο τρίτος πυλώνας, μέχρι Δευτέρα βράδυ βέβαια τρίτος πυλώνας. Υπήρχε ένα νομοθετικό σώμα και υπήρχε και ένα νομοθετικό σώμα στην νομοθετική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία που ήδη υφίσταται, θα πρέπει να εξετάσουμε κάθε ξεχωριστό μέσο, εργαλείο, και να εξετάσουμε αν θα προταθεί αναθεώρησή του ή η αντικατασταση του από οδηγία. Σε περίπτωση που έχει δρομολογηθεί ήδη κάποια κατάσταση, θα πρέπει να εξετάσουμε ποιες προτάσεις θα πρέπει να επαναεξεταστούν στα πλαίσια της νέας νομοθεσίας, στα πλαίσια μιας οδηγίας. Ο τρίτος πυλώνας, όπως λέω συνήθως, έχει εξαφανιστεί σε μεγάλο βαθμό. Φυσικά αυτό που πλέον μπορούμε να αποκαλέσουμε ο πρώην τρίτος πυλώνας είναι πολύ σημαντικός γιατί περιλαμβάνει νομικούς ορισμούς, γιατί υποκείται σε πολύ συγκεκριμένους ε, κανόνες από τη συνθήκη σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την Δανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι όμως αποκλειστικά τα μέλη αυτά, λόγω μηχανισμών που περιλαμβάνονται. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να ορίζουμε τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία στον ε, ποινικό τομέα, τον, πρώτο, τον τρίτο πυλώνα δηλαδή, ιδάλλως, γιατί είναι πολύ σημαντική, σημαντικό το περιεχόμενο. Θα υπάρξει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση Omnibus για το Γενικό Νόμο. Θα σας την κοινοποιήσουμε σήμερα το απόγευμα και προετοιμάζεται φυσικά εδώ και καιρό λόγω της θέσης ισχύ της ε, Συνθήκη της Λισαβόνας θα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να αντικατασταθούν οι νομοθεσίες στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα εν ευθέτω χρόνο. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πότε θα εξαρτηθεί από τους νέους επιτρόπους. Θα τους συναντήσετε άλλωστε και στις ακροάσεις. Θα τους θέσετε σχετικά ερωτήματα φαντάζομαι. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Θέλει κανείς ε, συνάδελφος να πάρει το λόγο. Ήσασταν πολύ πιστικός. Μεγάλη διαφορά με πριν που σας βομβαρδίσαμε με ερωτήσεις. για την ε, Επιτροπή του άρθρου 29. Είχαμε την αίσθηση χτες ότι χρειάζεται πιο πολύ υποστήριξη, γιατί είναι συμβουλευτικό σώμα και θα διαδραματίσει όλο ένα και πιο σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της νέας συνθήκης. Δεν αρκεί να περιμένουμε να διαμορφωθεί πλήρως το νέο πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων. Αλλά είπατε... Ναι, ναι, ναι, δεν είμαι... Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τον προϋπολογισμό, όντως, δίκιο έχετε. Αλλά ίσως να είναι και ένα θέμα το οποίο μπορούμε να θέσουμε προς τους υποψήφιους ε, επιτρόπους κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, γιατί είναι επιλογή πολιτική ουσιαστικά, πώς οργανώνουμε τη γραμματεία μας, που αφιερώνουμε τα κονδύλια μας και νομίζω ότι θα πρέπει να ρωτήσουμε τους επιτρόπους κατά πόσο προτίθενται να υποστηρίξουν περαιτέρω την ομάδα εργασίας. Μάλιστα, Νομίζω ότι συνάδελφοι έτσι ολοκληρώνουμε την σημερινή μας συνεδρίαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ νέου τον κύριο Φούλ για τον χρόνο που μας αφιέρωσε. Έχουμε στο, στις 12 προβλέπεται συνεδρίαση των συντονιστών, προς το παρόν όμως ε, λίγη συνεδρίαση.